Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Καταρχήν, να καλωσορίσουμε ένθερμα, ιδιαίτερα ένθερμα, την κυρία Ρέντινγκ και να δεν αστείευουμε. Σήμερα το πρωί σε αυτή την αίθουσα έκανε κρύο, πολικό ψύχος. Και τώρα μάλλον βιώνουμε ένα σοκ θερμοκρασίας, γιατί από το πολικό ψύχος τώρα νομίζω ότι υδρώνουμε και μας επιβλήθηκε αυτή η υπερθέρμανση. Έτσι λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω που μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό, σας παρακαλώ ξανασκεφτείτε το. Γιατί μιλάμε εδώ για δραστική άνοδο της θερμοκρασίας. Νομίζω ότι κάτι διάμεσο πρέπει να υπάρχει δηλαδή από το πολικό ψύχος ε, σε αυτές τις ε, υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, ας περάσουμε στις εργασίες μας. Αφού καλωσόρισα την Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων, για την ενδιάμεση αναθεώρηση του προγράμματος Στοκόλμης. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ολοκληρώνεται η σκληρή εργασία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για το 2012 σε σχέση με την αναθεώρηση του προγράμματος της Στοκχόλμης, γιατί μας υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα της Στοκόλμης ιδρύθηκε από τη Σουηδική Προεδρία όταν τέθηκε σε ισχύ η ίδια συνθήκη της Λισαβόνας Δηλαδή αφορά ουσιαστικά μια ευρωπαϊκή πολιτική, ο χώρος ελευθερίας δικαιοσύνης και ασφάλειας και φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης μέσω της ε, τακτικής νομοθετικής διαδικασίας για τους περισσότερους φακέλους με τις οποίες ασχοληθήκαμε για να προσδώσουμε περιεχόμενο στο χώρο ελευθερίας δικαιοσύνης και ασφάλειας. Έτσι λοιπόν, τρία έτη μετά, αφού τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, αξιολογούμε την κατάσταση και θα έχουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας για την ίδια συνεθεώρηση του προγράμματος Στοκόλμη και εγώ διορίστηκα εισηγητής ε, από την Επιτροπή Λίβη. Καλωσορίζουμε και τα μέλη των Επιτροπών Νομικών Θεμάτων και στεγματικών Υποθέσεων για αυτή την ανταλλαγή απόψεων που θα λάβει χώρα αφού θα ακούσουμε την παρουσίαση της κυρίας Ρέντινγκ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Uh, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τις επιτροπές μας έδωσαν τη δυνατότητα σήμερα να σας πούμε τι κάναμε με το πρόγραμμα αυτό. Γιατί είναι ωραία όταν είναι γραμμένα στα χαρτιά τα προγράμματα, αλλά μπορούν και να συζητηθούν. Πάνω απ' όλα αυτό που μετράει όμως και το είπε καθαρά ο πρόεδρος είναι από ένα πρόγραμμα να βγει δράση και αυτό προσπάθησα να κάνω αφού του ανέλαβα αυτή την ευθύνη. Θυμάστε ακόμα την πρώτη μας συζήτηση για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Οι απόψεις διήσταντο. Κάποιοι έλεγαν ότι είναι εξαιρετικό, άλλοι έλεγαν ότι είναι αρκετά καλό, αλλά οι περισσότεροι συμφωνούσαν ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης θα είναι ένα εργαλείο για να μας βοηθήσει να γίνει ο χώρος της δικαιοσύνης πραγματικότητα. Ένας οδικός χάρτης, ο οποίος άνοιγε νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Κοινοβούλιο θα γινόταν ε, πραγματικός συνομοθέτης μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσετε ότι διανύσαμε πολύ δρόμο οικοδομώντας αυτόν τον ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης και ότι επιτελέσαμε πρόοδο επί σειρά θεμάτων, ε, δικαιοσύνη για την ανάπτυξη που δεν υπήρχε, τη δημιουργήσαμε, ποινική νομοθεσία, θεμελιώδη δικαιώματα, ισότητα, ε, πολιτική κατά των διακρίσεων, όλα αυτά ήταν στην ημερήσια διάταξη και έγιναν πολλές βελτιώσεις. Και όλες αυτές οι βελτιώσεις νομίζω ότι κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών. Το πρώτο στοιχείο βέβαια που πρέπει να δούμε είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα δικαιοσύνης αξιόπιστο και αποτελεσματικό γιατί αυτό περιμένει ο κόσμος από μας. Ο κοινό ευρωπαϊκός νόμος για τις πωλήσει επιχειρήσεις για την ανάπτυξη, να μειώσουμε τα εμπόδια για το διασυνοριακό εμπόδιο, να γίνονται αγορές με ασφάλεια σε όλα τα κράτη-μέλη, με ασφάλεια για τους καταναλωτές, επέκταση σε νέες αγορές στην Ευρώπη χωρίς υπερβολικό νομικό κόστος για τις επιχειρήσεις, ε, οπότε αυτά όλα είναι, ε, ετοιμάζονται. Και όπως είδα και οι συζητήσεις για όλα αυτά στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξελίσσονται προς τη σωστή κατεύθυνση και καλά. Η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, θυμάμαι όταν το συζητήσαμε, ε, είμαστε πολύ στριμωγμένοι και καταφέραμε να το βάλουμε πάλι σε τροχιά για να συζητηθεί και θα εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη μέχρι τον Ιούνιο του 2014. Μεταξύ άλλων θα είναι πολύ σημαντικό για τις επιγραμμικές ε, αγορές. Ένα άλλο θέμα είναι οι διαδικασίες ε, διασυνοριακών διαφορών για να πάρουν τα χρήματα που τους οφείλουν και οι ε, οφειλέτες δεν θα κρύβονται σε άλλο κράτος μέλος, δεν θα μπορούν πια για να μην πληρώνουν μετά η μεταρρύθμιση των Βρυξελών 1 όπου σταματήσαμε τη διαδικασία εξεκουάτουρ της κήρυξης εκτελεστότητας, πράγμα που θα εξοικονομήσει χρήματα για όλους, γιατί οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε μια χώρα μέλος αυτομάτως θα αναγνωρίζονται και σε άλλο κράτος μέλος και σε αυτή τη λογική του ανοίγματο των συνόρων για να διευκολυνθεί το εμπόριο σε ειδικέ αγορές για τις μικρές, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ε, καταναλωτές. Το νέο πακέτο για την αφαιρεγγιότητα που το παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα και που αλλάζει την άποψη για την αφαιρεγγιότητα. Ε, όταν κάποια εταιρεία πτώχευε, έπρεπε, θα έπρεπε να διαλυθεί η εταιρεία για να πληρωθούν οι πιστωτές. Και αυτό σε τελευταία ανάλυση σήμαινε απώλεια θέσεων εργασίας. Το νέο πακέτο αφαιρεγγιότητας ε, προσπαθεί να βρει τρόπους ε, ώστε οι βιώσιμες επιχειρήσεις να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία και να διασώζονται οι θέσεις εργασίας. Είναι δηλαδή τελείως διαφορετική προσέγγιση της πτώχευσης. Μετά, οι γυναίκες σε Συμβουλή Επιχειρήσεων, εκτός από το θέμα των δικαιωμάτων, υπάρχει και το θέμα της ανάπτυξης. Έχουμε δει ότι οι εταιρείε με γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτό απαντά και στις ελλείψεις ειδικοτήτων στην Ευρώπη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια πια στην Ευρώπη να μην αξιοποιούμε τα γυναικεία προσόντα και ειδικότητε όπως θα έπρεπε. Τέλος, αλλά πολύ σημαντικό, η μεγάλη μεταρρύθμιση στην προστασία των δεδομένων, που είναι μια από τις μεταρρυθμίσεις και πάλι, που είναι διπλού χαρακτήρα. Πρώτον, έχουμε καλύτερη προστασία των ε, δικαιωμάτων κάθε ατόμου, ε, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και από την άλλη έχουμε άνοιγμα της ε, αγοράς για τις εταιρείε και αντί να έχουμε 27 συγκρουόμενους κανόνες έχουμε έναν κανόνα. Οπότε μειώνουμε το φόρτο για τις επιχειρήσεις και αυξάνουμε και το επίπεδο της προστασίας για τον κόσμο και μειώνουμε το φόρτο για τις επιχειρήσεις. Οι δύο προτάσεις που δημιουργούν το πακέτο συζητήθηκαν πολλές φορές στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, διορθώσουμε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει γενικότερα θετική προσέγγιση, δέσμευση ε, υπέρ όλων αυτών. Οπότε οι εργασίες εξελίσσονται πολύ καλά και η Ιρλανδική Προεδρία θέλει το θέμα αυτό να το βάλει ανάμεσα στις προτεραιότητές της στο επόμενο εξάμεινο. Οικογενειακό δίκαιο. Εδώ ε, πάλι ε, ήταν ένας τομέας τον οποίο δεν είχαμε αγγίξει στο παρελθόν γιατί εδώ ήταν 100% θέμα επικουρικότητας. Προχωρήσαμε πολύ καλά και ταχύτατα. Ναι, οι κανόνες για το διαζύγιο και τη νομική διάσταση ε, μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας. Η πρώτη ενισχυμένη συνεργασία στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμάστε, που επιτρέπει στα ζευγάρια να διαλέγουν ε, το, ή τη διάσταση ή το διαζύγιο πιο δίκαιο, ποιας χώρας θα, το, θα τα διέπει. Και το ίδιο και για την διαδοχή, την κληρονομία. Επίσης, στην ποινική νομοθεσία έχουμε θέσει κοινά πρότυπα για δίκες, δίκες σε όλη την επικράτεια της Ένωσης, ελάχιστους κανόνες, ώστε κάθε πολίτης να ξέρει ότι όπου και να ταξιδέψει θα έχει τα ελάχιστα αυτά δικαιώματα, αν συμβεί κάτι. Ο δικός χάρτης για τα δικονομικά δικαιώματα, το δικαίωμα για τη μετάφραση, για τη διερμηνία, το δικαίωμα για την ενημέρωση σε ποινικέ υποθέσεις, διαδικασίες και προχωρούμε και στο πιο σημαντικό δικαίωμα να διασφαλίσουμε την πρόσβαση σε δικηγόρο, συνήγορο που είναι σημαντικό για μια δίκαιη δίκη. Μαζί με σας και εγώ είμαι πολύ περήφανη, διότι δεν είδαμε μόνο τις ε, παραδοσιακές ποινικέ διαδικασίες, αλλά βάλαμε το θύμα στο επίκεντρο, στην καρδιά του συστήματος δικαιοσύνης. Έχουμε την οδικία για τα θύματα που ήταν πραγματικό ρηξικέλευθο βήμα. Επίσης η εντολή ποινική προστασίας αποφασίστηκε, η εντολή ένταλμα ε, αστικής προστασίας επίσης ε, τώρα θα είναι έτοιμη πολύ γρήγορα, ετοιμάζεται μαζί με μια οδηγία για ε, διασυνοριακή προστασία θυμάτων βίας κυρίως γυναίκες είναι αυτά τα θύματα, όλα αυτά σημαίνουν ότι θα έχουμε ένα προστατευτικό περιβάλλον για τις γυναίκες αυτές. Και ξέρω ότι θέλετε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις ε, σε αυτό το θέμα πολιτικής προστασίας, ε, ε, αστικής προστασίας ποινική και αστική. Και όταν μιλώ για θύματα, βέβαια, δεν μιλώ μόνο για τι γυναίκε, μιλώ και για τα παιδιά, τα οποία πάντα ήταν προτεραιότητα στην κοινή μα εργασία. Η οδηγία για τα θύματα έχει ιδιαίτερες διασφαλίσεις για τα παιδιά. Ε, υιοθετήθηκε το 2011 είναι για την καταπολέμηση της σεξουαλικής ε, κακοποίησης, παιδικής πορνογραφίας και αυτά ε, ενισχύουν ε, το σύστημα προστασίας για τα παιδιά και της δίωξης των ε, ενόχων και μην ξεχνάτε και την ατζέντα της Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού του, από τον Ιανουάριο του 2011 για να δούμε σε προοπτική τα δικαιώματα των παιδιών ε, τα οποία ε, θεσπίζονται στον χάρτη και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Έχουμε λοιπόν ε, οικοδομήσει πάνω στα θεμελιώδη δικαιώματα όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά και με νομοθετήματα. Θα πρέπει όλα αυτά να είναι συνεπή προς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την νομοθεσία της Ευρώπης. Τον Οκτώβριο του 2010 θα θυμάστε τη στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή του χάρτη ε, είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα την περασμένη εβδομάδα στα πλαίσια της έκθεσης της κυρίας Φλασίκοβα Μπένοβα. Ο χάρτης ε, δίνει το μέτρο που θα τα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι ο χάρτης θα την χάνει σεβασμού όπως έλεγχος ε, συμμόρφωσης ε, της νέας νομοθεσίας με το χάρτη. Επίσης, ε, ο κατάλογος των θεμελιωδών δικαιωμάτων που εφαρμόσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τρόπο οριζόντιο για όλες τις νομοθεσίες και χαίρομαι διότι και το Συμβούλιο εφαρμόζει τώρα αυτόν τον κατάλογο όταν εξετάζει τις τροπολογίες που θα προτείνει επί των κειμένων μας. Και επίσης υπάρχει και η ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του χάρτη που δημοσιεύτηκε για δεύτερη φορά. Περνώ σε ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο επεξεργάζομαι με συναδέλφους σοβαρές προσπάθειες για την καλύτερη ε, κα, ε, καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος προσπαθήσαμε να ε, χτυπήσουμε στον τραπεζικό τομέα ε, καταχρηστικές πρακτικές. Ε, επίσης η οδηγία κατά της απάτης που στοχεύει στην εναρμόνιση των κανόνων των κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης. Η πρότασή μας περιλαμβάνει και κοινέ ελάχιστες κυρώσεις για την αποτροπή των απαταιώνων. Και Ακολουθεί μία ανακοίνωση και μία έκθεση για θέμητες εμπορικές πρακτικές. Ε, πρόκειται για οδηγίες για αυτό το θέμα που στις αρχές του επομένου έτους θα υποβληθούν και σε εσά και θα ενισχύσει την επιβολή του νόμου ε, όχι μόνο σε τομείς όπως επιγραμμικές αγορές και μεταφορές. Δουλεύουμε επίσης και σε ε, έγγραφα αστικού δικαίου για να με εμπόδια σε πολίτες που θέλουν να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους της ελεύθερης διακίνησης. Ε, επίσης ε, χειρίζομαι ένα δύσκολο θέμα που είναι μια αναθεώρηση της οδηγίας ε, για τα ταξίδια που λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές στην αγορά. Διότι όταν καταρτήσαμε πρώτη φορά την οδηγία αυτή δεν υπήρχαν χαμηλού κόστους μεταφορής, ούτε ε, κρατήσεις μέσω διαδικτύου. Πρέπει λοιπόν η νομοθεσία μας να προσαρμοστεί για να λάβει υπόψη τις αλλαγές στην αγορά και τις αλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών. Είμαι βέβαιη ότι πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε θα μπορέσουμε να προσθέσουμε και άλλα ακόμη επιτεύγματα στον κατάλογο αυτό γιατί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο διαπραγματεύονται και προχωρούν καλά σε σχέση με τα, τη διάσταση και το διαζύγιο και την επίπτωση στην περιουσία και την προξενική προστασία ε, των πολιτών που έχουν δυσκολίες όταν ταξιδέψουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή είδαμε σε κάποια κράτη-μέλη να υπάρχουν δυσκολίες και είδαμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ένα καλά λειτουργικό ε, αστικό σύστημα και εμπορικό σύστημα, ούτως ώστε να υπάρχει ε, ασφάλεια δικαίου για τους επενδυτές. Γιατί αν δεν υπάρχει η νομική ασφάλεια, δεν πρόκειται να επενδύσουν οι ενδιαφερόμενοι. Γι' αυτό και έκανα τη σχετική πρόταση στο Κοινοβούλιο, όταν κάναμε στην Ολομέλεια μια πολύ δύσκολη συζήτηση. Τώρα έχουμε συμπεριλάβει στην ε, διαδικασία μας αξιολόγησης της εξέλιξης των οικονομιών και των προϋπολογισμών των κρατών μελών ένα βαθμολόγιο των επιδόσεων των κρατών μελών για να δούμε Πώς λειτουργεί το σύστημα δικαιοσύνης. Η ανεξαρτησία της ε, δικαστικής εξουσίας είναι πολύ σημαντικό θέμα, όπως επίσης και ε, η η, η, η, συμφόρηση στις υποθέσεις που συσσωρεύονται για να αποφασιστούν. Στις 27 Νοεμβρίου υπέβαλα μια ανακοίνωση για την, ε, για την οδηγία για την παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση για να έχουμε καλύτερη διασυνοριακή εφαρμογή της οδηγίας χρειάζεται να στοχεύσουμε ειδικού προβληματικούς τομείς ε, τα πάτες με καταλόγους ε, για, τους οποίους, τις οποίες είχατε και εσείς κάνει καταγγελίες και το 2013 προβλέπονται μέτρα ε, καταπολέμησης και για να ε, είμαστε ικανοποιημένοι και ο πρόεδρος σας και εγώ πρέπει να σας πω ότι το γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα είναι στο στόχαστρό μας και θα βάλουμε τώρα θα, θα υποβάλουμε πρόταση το 2013. Το γραφείο αυτό θα αντιμετωπίζει θέματα ε, που αφορούν αδικήματα και εγκλήματα ε, ενάντια στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να μεταρρυθμίσουμε και την Eurojust σε αυτά τα πλαίσια για να είναι πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος και για να επικουρούν και τα κράτη-μέλη στην καθημερινή του συνεργασία. Με αυτή την ευκαιρία ε, θα εργαστώ και για την Eurojust και τον, ε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ε, και θέλω να πω ότι η Κομισιόν έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τις δραστηριότητες της Eurojust και μπορεί και να συμμετέχει, να συμμετέχει στη διαδικασία δημιουργίας του Γραφείου του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Και για τα δικονομικά δικαιώματα είμαστε βέβαια στο μέσον της οδού, δεν έχουμε ε, τελειώσει. Θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω στην υπόθεση της αθωότητας, να έχουμε ιδιαίτερες διασφαλίσεις για ευάλωτα πρόσωπα, όπως ανακοίνωσα και στα πλαίσια του πακέτου για τα θύματα και η νομική βοήθεια. Όλα αυτά θα τα εντάξω σε ένα πακέτο και θα τα πάρετε θα πάρετε την πρόταση το δεύτερο εξάμεινο του 2013. Όλοι γνωρίζουμε ότι ένα από τα στοιχεία της αμοιβαία εμπιστοσύνης, χωρίς την οποία η αμοιβαία αναγνώριση και η συνεργασία ε, των, ε, της δικαιοσύνης δεν μπορεί να λειτουργήσει, στηρίζεται μεταξύ άλλων ε, και στο σύστημα της κράτησης. Θέλουμε να έχουμε κοινωνική αποκατάσταση, και να μειώσουμε ε, την προφυλάκηση. Ε, θέλουμε μια στρατηγική για να διασφαλίσουμε ότι οι τρεις ε, αποφάσεις πλαίσιο για την, κράτηση θα εφαρμόζονται σωστά από τα κράτη-μέλη μέχρι το, δύο, το τέλος του 2014. Γνωρίζετε ότι για τις αποφάσεις πλαίσιο δεν μπορεί να υπάρχει άμεση παρέμβαση ούτε της Κομισιόν, ούτε του Κοινοβουλίου, ούτε του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου γιατί είναι πριν από, το, από τη Λισαβόνα. Όμως είναι σημαντικό το πλαίσιο για τις κρατήσεις να εφαρμόζεται, γιατί αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε μεγάλες αντιδράσεις από κάποια δικαιικά συστήματα ε, προκειμένου περί απελάσεων, εκδόσεων. Το τέλος για την πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα ε, πρέπει να συνάδει με το Ευρωπαϊκό Σύστημα ε, Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας και το Συμβούλιο εξετάζει κάποιες λεπτομέρειες ε, ενω ενώ κάνα δύο κράτη-μέλη δημιουργούν προβλήματα, αλλά είναι σημαντικό να προχωρήσουμε γρήγορα προς την κατεύθυνση μιας ταχείας προσχώρησης. Και ένα τελευταίο στοιχείο, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η προπαρασκευαστική μας δουλειά για την Ευρώπη, για τους πολίτες, ε, προχωρεί ολοταχώς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ήταν πολύ θετικό απέναντι στις δραστηριότητες που είχαμε μέχρι τώρα, συνεδριάσεις στο Δημαρχείο και φαντάζομαι ότι το 2014 οι βουλευτές θα δραστηριοποιηθούν πολλοί συμμετέχοντας σε δημόσιες εκδηλώσεις για να ακούσουν τι έχουν να πούν οι πολίτες. Κύριε Πρόεδρε, αυτά ήταν και αυτό ήταν μια πολύ μικρή σύντομη περίληψη. Ε, είδατε ότι ασχοληθήκαμε με πολλές δράσεις, δουλέψαμε ταχύτατα και όλα αυτά δεν θα ήταν, δεν θα δυνατό να γίνουν αν δεν είχε κάνει τη δική του δουλειά το Κοινοβούλιο και την έκανε καλά και σας ευχαριστώ όλους. Και πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές που πραγματικά ήταν μεγάλη βοήθεια και μπόρεσαν να προχωρήσουν το χώρο της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε, ευχαριστώ Αντιπρόεδρε Ρέντινγκ για την παρουσία παρουσίαση όλης καταστάσεως όσον αφορά το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Γεννήθηκε και επιμένω γι' αυτό την ίδια στιγμή θέση σε ισχύ της συνθήκης της σαν κρίσιμο συστατικό στοιχείο της συνταγματικής μεταρρύθμισης που έλαβε χώρα με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Άλλαξε η φύση του χώρου ελευθερίας δικαιοσύνης ε, και ασφαλείας. Τρία χρόνια πέρασαν. Τρία χρόνια. Ακριβώς τρία χρόνια. Και πρέπει να παραδεχτούμε επίσης τις πρωτοβουλίες που αναλήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σημειώθηκε έτσι ουσιαστική πρόοδος σε θέματα που μας απασχολούν. Θέματα που αγαπάει η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, όπως είναι το πακέτο για τα δικονομικά δικαιώματα και το πακέτο για την προστασία των δεδομένων. Και οι δύο πρωτοβουλίες μας αφορούν. Και πριν παρουσιάσω τον κατάλογο των μελών που θέλουν να μιλήσουν, να πω κάτι κι εγώ, ως εισηγητής επιφορτισμένος με την ενδιάμεση αναθεώρηση που είναι ε, πρωτοβουλία της Επιτροπής μας των Πολιτικών Ελευθεριών. Θα ήθελα να τονίσω λοιπόν το πόσο σημαντικό είναι το χρονοδιάγραμμα. διότι είναι το τέλος του 2012 και πλησιάζουμε το 2013 που θα είναι ο τελευταίος πλήρης χρόνος της θητείας αυτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά τώρα περισσότερο από ποτέ αν θέλουμε να πετύχουμε τα ευκταία αποτελέσματα διότι αν δεν τα καταφέρουμε το 2013 Υπάρχουν ελάχιστε πιθανότητες να δει το θέμα αυτό πριν το τέλος της θητείας μας. Σίγουρα πρώτους μήνες του 2014 θα ξαναξεκινήσουμε προεκλογική εκστρατεία, θα είμαστε καθοδόν προς τις εκλογές, οπότε πρέπει να έχουμε υπόψη μας πόσο σημαντικό είναι το χρονοδιάγραμμα. Γι' αυτό εξετίμησα την αφοσίωσή σας, ούτως ώστε εγκαίρως να τα πετύχετε όλα αυτά και είπατε συγκεκριμένα ότι συμπεριλάβατε και το, την υπηρεσία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Υπηρεσίας, για να γίνουμε αποτελεσματικότεροι στην αντιμετώπιση διασυνοριακών σοβαρών εγκλημάτων. Σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου 83, που αναφέρεται σε ποινικά δικήματα διασυνοριακού χαρακτήρα. Και το άρθρο 86 που καθορίζει τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέο θεσμό, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Υπηρεσία, βάσει της εμπειρίας του Eurojust μέχρι τώρα. Άρα, είναι σημαντικό με βάση όλα αυτά να ασχοληθούμε με την εφαρμογή και τις παραβιάσεις. Μιλάμε για τα θεμελία, θεμελιώδη δικαιώματα που δεν είναι ευσεβείς πόθη πλέον. Έχουν την ίδια νομική αξία σαν, όπως και οι ίδιες οι συνθήκες, οι ίδιες οι συνθήκες Λισαβόνας. Έτσι θα πρέπει να ειδωθεί η Ευρωπαϊκή Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι θέμα κράτους δικαίου είναι θέμα δεσμευτικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επενούμε την πρότασή σας, συνεπώς για να υπάρξει, να θεσπιστεί ένα σύστημα βαθμολόγησης όσον αφορά το κατά πόσο γίνεται σεβαστό το κράτος δικαίου και πώς αυτό μας δείχνει πώς προχωράει όλη η προσπάθεια. Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη ότι είναι σημαντικό να υπάρξει συντονισμό μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Εδώ έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκπροσωπούμε 500 εκατομμύρια πολίτε συνολικά. Αυτό είναι το κοινοβούλιο που αντιπροσωπεύει την ευρωπαϊκή σφαίρα και το ευρωπαϊκό επίπεδο λήψη αποφάσεων και ευθυνών. Το κοινοβούλιο εκπροσωπεί, παγιώνει την εκπροσώπηση και τη δυνατότητα ελέγχου δραστηριότητας του πολιτικού τομέα. Κάτι που είναι καθαρά ευρωπαϊκό χαρακτηριστικό και γνωρίζουμε άριστα όμως ότι τα κράτη-μέλη πάντα είναι εκεί με εθνικά κοινοβούλια, το κάθε κράτος και τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να γίνονται σεβαστά. Να γίνονται σεβαστά όσον αφορά τη συμπλήρωση των προσπαθειών μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης να γίνονται γνωστές οι νομοθετικές αρμοδιότητες των κρατών μελών σε ευαίσθητα θέματα, όπως του οικογενειακού δικαίου, όπως κάποιων τομέων του ποινικού δικαίου. Θα πρέπει να είμαστε πιο πρόθυμοι να συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά. Γνωρίζουμε ότι μιλάμε για ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό το Ευρωκοινοβούλιο έχει καθήκον να γίνεται ένα και πιο ψηλό, να υψώνει το ανάστημά του και να γεμίζει το χώρο με την παρουσία του. Δεν πρέπει να υποχωρούμε. Δεν πρέπει να θα τα δικά μας περιθώρια λιγμών. Πρέπει να γεμίζουμε το χώρο μας με περιεχόμενο. Αλλά χρειάζεται και άλλη προσπάθεια συνεργασίας την άνοιξη του 2013 να ετοιμαστεί μια νέα διακοινοβουλευτική διάσκεψη με συμμετοχή Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου συνεργαζόμενοι αυτοί οι φορείς θα εποπτεύουν την όλη εφαρμογή της συνθήκης της και κυρίως όσον αφορά τα θεμελιώδη ε, δικαιώματα. Επιμένω από αυτού. Ε, διατηνόμεθα ότι είμαστε απαιτητικοί όσον αφορά τις χώρες που θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χτυπάνε την πόρτα. Κρούν τη θύρα. Και κατά πόσο είναι αποτελεσματικά την κριτήρια της για το κράτος δικείου, θεμελιώδη, δικαιώματα, όλα αυτά. Όταν είμαστε απαιτητικοί για όλα αυτά, για τα υποψήφια κράτη-μέλη, θα πρέπει να είμαστε απαιτητικοί και για τα ήδη υπάρχοντα μέλη. Αυτές οι αρχές να μην είναι λιγότερα αποτελεσματές από τη στιγμή που χώρες γίνονται πλήρη μέλη της λέσχης, από ό,τι ήταν πριν όταν ήθελαν να μπουν στη λέσχη και έκρουαν τη θύρα και προσπαθούσαν να θέσουν το πόδι τους στην πόρτα και να μπουν στη λέσχη. Πρέπει να επαγρυπνούμε για να μην μειώνεται την επόμενη μέρα η αποτελεσματικότητα των αρχών αυτών. Τούτων λεχθέντων εκφράζω την πρόθεσή μου μήνα Ιανουάριο, αρχή, τέλος Ιανουαρίου να σας δώσω ένα πρωτόλιο της ενδιάμεσης Έκθεση εκ μέρου Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών για συνεργασία με επιτροπέ. και λέγοντας αυτό ξεκινάω το μέλη. Η κυρία Ματιέ. Έχετε το λόγο κυρία Ματιέ. Ευχαριστώ. Καταρχήν ευχαριστήσω την κυρία Ρεντίνκ που ήρθε εδώ στην ε, παρουσίασή μα καθώς πρόκειται για την ε, τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Λιμπή για φέτος. Ε, σας ευχαριστώ για όλες τις προτάσεις της Κομισιόν, ε, κυρίως για το πρόγραμμα Στοχόλμης. Όταν σας ακούμε και όταν βλέπουμε όλες τις προτάσεις της Κομισιόν, συνειδητοποιούμε ότι έχουμε προχωρήσει πολύ από την έναρξη της θητείας και αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί πραγματικά υπήρχε ένα κενό σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δικαιοσύνη και αρχίζει να καλύπτεται τώρα αυτό το κενό. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε ικανοποιημένοι με τι προτάσει που έχετε υποβάλει και με το έργο του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό το τομέα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι πρέπει να γίνει και άλλη δουλειά και ιδίω ήθελα να σα ρωτήσω, παραδείγματο χάρη, ε, αυτή τη στιγμή μιλάμε για την οδηγία για τους νομικούς ε, ουσιαστικά το έχετε συνδέσει αυτό την ε, νομοθεσία για τη δικαιοδοσία με την οδηγία για τους δικηγόρους και έχετε κάποια πρόταση για το μέλλον και επίσης σε ό,τι αφορά ε, την οδηγία για την διερμηνία. Λείπουν κάποιοι πόροι συχνά στα κράτη-μέλη προκειμένου να μπορεί να δίδεται αποτελεσματικά η διερμηνία, να παρέχεται αποτελεσματικά η διερμηνία. Έχω ένα παράδειγμα, ε, θα γνωρίσετε στο Βέλγιο ότι είναι Λήφθη ένας Βραζιλιάνος με τέσσερα κιλά κοκαίνης και δεν μπορούσαν να βρουν κάποιο διερμηνέα για τα πορτογαλικά, ακόμη και αν βρισκόμαστε στο Βέλγιο. Και Έχουμε, ξέρετε, αρκετού διερμηνείς ε, στα κράτη-μέλη και επειδή δεν υπήρχε διερμηνέας άφησαν ε, να φύγει αυτός ο Βραζιλιάνο, να επιστρέψει στην πατρίδα του γιατί ε, δεν έγινε σεβαστή ο νόμο, εσεί σκοπεύετε να συστήσετε κάποιο μέσο ακριβώς για να καολύψετε αυτή την αδυναμία των κρατών μελών σε αυτό το πλαίσιο. Επίσης, σε σχέση με τη διαφθορά, Γνωρίζετε ότι σε κάποια κράτη-μέλη και στη Γαλλία μας δακτυλοδείχνουν ε, γιατί δεν ε, καταπολεμάτε παρκώς η διαφθορά. Έχετε την πρόθεση να υποβάλλετε κάποια πρόταση για να ε, προστατεύσετε όσους προβαίνουν σε καταγγελίες, τους whistleblowers. Και να θέσω και μια ακόμη ερώτηση. Μιλήσατε για τον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα. Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής, ποιο θα ήταν το πεδίο εφαρμογή ε, για τον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα, ε, πέρα από το να προστατεύει τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχετε την πρόθεση να διευρυνθούν οι αρμοδιότητές του, να καλύπτεται δηλαδή και το οργανωμένο έγκλημα και να έχει και άλλε αρμοδιότητε. Αυτά από μένα. Θα αφήσω το λόγο στους υπόλοιπου συναδέλφους. Η κυρία Φαγιόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Μισό λεπτό να... Θα μιλήσω στα σλοβενικά, διότι υπάρχει διερμηνία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που βρήκατε χρόνο να έρθετε, ενώ πολλοί συνάδελφοι δεν είναι πια εδώ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση, την ενημέρωση και το έργο σας. Θέλω να μιλήσω για κάτι που δεν αναφέρθηκε, αλλά είναι πολύ σημαντικό και αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από λίγο καιρό ε, ψηφίσαμε με μεγάλη πλειοψηφία μια έκθεση και ένα ψήφισμα για την CIA δεν πρόκειται για νέες διαπιστώσεις, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με σοβαρές παραδιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί του εδάφους της Ένωσης και καλέσαμε την Κομισιόν να ε, διερευνήσει τι γίνεται στα κράτη-μέλη και να λάβει μέτρα που θα διασφαλίζουν ε, καλύτερες, αποτελεσματικότερες έρευνες και θα αναλαμβάνουν την ευθύνη για αυτές. Εμείς στην Ευρώπη δεν μπορούμε να απευθύνουμε, ε, κλίση, να απευθύνουμε για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να καταδικάζουμε τις αραβικές χώρες και να αγνοούμε τι γίνεται σε εμά. Την τελευταία, την περασμένη εβδομάδα έγινε μια έκθεση για τη Μακεδονία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο διαπιστώνει ότι το αρμόδιο δικαστήριο εκεί δεν άρχισε ε, σωστές διαδικασίες και έρευνες. Πρέπει να πω ότι ανησυχώ πάρα πολύ και αγανακτώ κιόλας για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις τελευταίες μέρες του χρόνου ε, η οποία πρέπει επίσημα να ε, αντιδράσει ε, στις, στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου και στις εκθέσεις και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι πάρα πολλές επίσης οι εκθέσεις των δημοσιογράφων. Υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που απεφάνθηκε αυτό. Θέλω λοιπόν να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το τελευταίο ψήφισμά μας θα το λάβει υπόψη της θα αντιδράσει ε, στις αναφορές σχετικά με τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ντάφ. Καλώς σας απόγευμα, κυρία Ρέντινγκ. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Επιτροπή θα παρουσιάσει προτάσεις για να ενδυναμώσει τις αρμοδιότητες ε, του Ευρωπαίου Εισαγγελέα σε σχέση με την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού εγκλήματος. Μπορείτε να μας πείτε αν έχετε ήδη ξεκινήσει να συζητάτε με την Βρετανική κυβέρνηση την προσέγγισή της για το αν θα συμμετέχουν ή θα αποκλειστούν από την πρόταση αυτή. Και μιλώντας ευρύτερα, πώς θα μπορούσατε να μας πείτε. Πόσο προβληματικά είναι τα opt-out που έχει πετύχει το Ηνωμένο Βασίλειο στην προσέγγιση του. στον τομέα δικαιοσύνης και ιστορικών υποθέσεων. Πόσα προβλήματα θέτουν αυτά τα opt-out στην πράξη για την Κομισιόν. Και με αφορμή αυτό, μήπως είναι πολύ νωρίς να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για την επόμενη μεταρρυθμίση της συνθήκης. Εγχείρημα που νομίζω ότι θα ξεκινήσει την άνοιξη του 2015. Ο πρόεδρος Μπαρόσο είπε ότι πρόκειται να δημοσιεύσει τις προτάσεις του, τις προτάσεις της Κομισιόν, για την άνοιξη του 2014. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πολύ αργά. Γιατί αν επιθυμεί να επηρεάσει την προεκλογική εκστρατεία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό της Κομισιόν για αυτά τα θέματα. Ήδη του χρόνου το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο του 2013 δηλαδή. Μπορείτε να μας πείτε αν η εμπειρία που έχετε μέχρι σήμερα από το πρόγραμμα της Στοκόλμης έχει προκαλέσει κάποιες σκέψεις για να υπάρξει αλλαγή στις αρμοδιότητες της Κομισιόν. στην κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ε, τμήμα της συνολικής δουλειάς σας σε αυτόν τον ε, ευαίσθητο πολιτικό τομέα. Ευχαριστούμε κύριε Ντεφ. κύριε Ντεφτίνη. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις. Κύριε Ρεντίνκα, αναφέρατε ότι στα μέσα του 2013 θα παρουσιάσετε μια ευρύτερη πρόταση, νομίζω το αποκαλείστε πακέτο, που θα συμπεριλαμβάνει και την νομική αρρωγή. Αυτά είναι καλά νέα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα το δούμε αυτό, αλλά μήπως μπορείτε να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες. Γιατί θα υπάρχει πακέτο και αν υπάρχουν νομοθετικές προτάσεις μέσα σε αυτό. Μιλάμε, έχουμε ξαναμιλήσει μάλλον για την ε, νομική αρρωγή, αλλά αν ε, θέλουμε να προωθήσουμε τη δικαστική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς να έχουμε ε, μια τέτοια νομική αρρωγή. Δηλαδή, δείτε τη συζήτηση για την πρόσβαση σε δικηγόρο και τη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και για την εντολή έρευνα, την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνα. Ε, αν δεν υπάρχει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πολίτε θα, μάλλον τα δικαιώματα των πολιτών ε, θα γίνουν σεβαστά και ότι θα βρουν το δίκιο τους. Θέλουμε λοιπόν κάποιες λεπτομέρειες από αυτό. Και κάτι ακόμα. Την περασμένη εβδομάδα στο Στραμβουργό συζητήσαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι αναφερθήκατε σε αυτό τον πίνακα αποτελεσμάτων ε, για τη δικαιοσύνη. Εγώ το θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Να σας ρωτήσω, είναι δυνατόν να διευρύνετε το πεδίο εφαρμογή, αλλά θέλω και να σας ρωτήσω Πότε θα δούμε πιο πρακτική πρόταση, δηλαδή τους δείκτες ε, για αυτόν τον πίνακα αποτελεσμάτων με τη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι ίσως ε, θα πρέπει να αρχίσουμε να προβαίνουμε σε μια σύγκριση της κατάστασης του σοβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άκουσα πριν και συνάδελφοι ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι και εμείς οι ίδιοι σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και ίσως να δακτυλοδείξουμε, να κατονομάσουμε και όλα στα κράτη-μέλη που δεν σέβονται τις ε, συμφωνίες ε, που έχουν συνάψει, που έχουμε συνάψει μεταξύ μας σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πότε λοιπόν ε, θα παρουσιαστούν αυτοί οι δείκτες για τον πίνακα αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ κύριο Σκύρκο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την Επίτροπο. Πληρέστατη η παράθεση των επιτευμάτων και του έργου. Τη συγχαίρω. Και αυτή και του συναδέλφους της. Έκαναν πολύ σκληρή δουλειά στα πλαίσια τη εντολή τους και τη αιτία του. Έχω μια ανησυχία όμως. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί γίνονται πάρα πολλά ταυτόχρονα, πάρα πολλά ζητήματα αντιμετωπίζονται στον τομέα αυτό πάντα αυξάνεται η ζήτηση και από πλευράς Κοινοβουλίου και από πλευράς της ίδια Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προκύπτει από γεγονότα που συμβαίνουν στα κάτι μέλη. Απαιτείται, υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για περισσότερες πράξεις. Να αντιμετωπίζονται περισσότερα ζητήματα. Με απασχολεί το θέμα της κρίσεως των επιτεγμάτων των ήδη επιτευχθέντων, πέρα από τα δρομολογηθέντα προγράμματα που συνεχίζονται. Και η Επίτροπος αναφέρθηκε στο σύστημα βαθμολόγησης στον τομέα της δικαιοσύνης. Και πάνω στα όσα είπε η κυρία Σαρτζεντίνη και εγώ θα ενδιαφερόμουν να δω ποιες παράμετροι, ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται για να γίνει η αξιολόγηση. Δηλαδή πώς βαθμολογείται κάθε, κάθε περίπτωση σαν πολιτικοί μπορούμε υποκειμενικά να κρίνουμε και να βαθμολογούμε. Είναι σαν διαγωνισμός ταλέντων, τύπου X Factor. Και ο καθένας κρίνει τι αποτελεί επιτυχία και τι όχι. Ποια είναι η φύση της διαδικασίας αξιολόγησης όσον αφορά το σύστημα βαθμολόγησης του τομέα της δικαιοσύνης. Και με ποιο τρόπο αξιολογούμε τα επιτευθέντα, πριν από χρόνια είχα συντάξει εγώ μια έκθεση για κοινέ ερευνητικές ομάδες. Γιατί υποστηρίζω ένθερμα την συνεργασία, την περαιτέρω που απαιτείται από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου στην Ευρώπη. Είχαμε σημαντικές επιτυχίες στον τομέα. Όμως, σε κοινέ ομάδες έρευνας δεν μπορώ να ξέρω επακριβώς πόσο επιτυχεί ήταν οι ομάδες, πόσο χρησιμοποιήθηκαν προς όφελο των Ευρωπαίων πολιτών και κάτι άλλο που θέλω να θίξω. Ε, το πώς εξελίσσεται το διαδίκτυο. Όλη μέρα θα μπορούσαμε να συζητούμε για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, για τις φρικτές καταχρήσεις που λαμβάνουν χώρα στο διαδίκτυο, κυρίως εκμετάλλευση παιδιών και γενικά γενική κλιματικότητα που έχει αναπτυχθεί στο διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί όλα αυτά να τα συναθρήσει σε μια συγκεκριμένη πολιτική για το διαδίκτυο, σε μια σαφέστερη προσέγγιση, γιατί πρόκειται περί διεθνού ζητήματο. Πώς ενδεχομένως θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε νομοθεσία, να δράσουμε για να αποφύγουμε αυτά τα φαινόμενα. Αυτοί που παρέχουν τις υπηρεσίες να, είναι, να λάβουν την, την ευθύνη για τα τεκτενόμενα. Διότι υπάρχει αρκετά αρνητική προσέγγιση και τυχαία που δεν προστατεύει τα παιδιά ούτε τον κόσμο καθόλου στην αναπτυσσόμενη αυτή τεχνολογία. Αυτά είχα να πω πρόεδρε και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζάροκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε. Κυρία Αντιπρόεδρε τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευχαριστώ για την πληρέστατη αυτή παρουσίαση που κάνατε. Για όσα έγινε το 2012, ευχαριστούμε την συνεργασία σας και προσβλέπουμε στην μελλοντική μας συνεργασία το 2013. Δύο ερωτήσει. Πρώτη, οι νομικέ πρωτοβουλίε σας. Και τώρα η αναθεώρηση τη οδηγία. Η τη οδηγία πώς θα πάει το 2013. Και πώς μπορεί να διαφέρει από την εκδοχή του 2007. Που ζητούσαμε, μάλλον επιβάλαμε κυρώσεις σε επιχάρτου. Επιβάλανε, ζητήσαμε από τις κυβερνήσεις να επιβάλλουν κυρώσεις και δεν το έκαναν οι χώρες. Άλλη ερώτηση. Κρίσιμο έτος το 2013 για την ένταξη των Ρωμά και τις ειδικές στρατηγικές. σε ποιο βαθμό μπορεί να κινηθεί και να αντιμετωπίσει τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτού και λαμβάνοντα υπόψη όλα αυτά που μας παρουσιάσατε. Ευχαριστώ κυρία Τζαρόκα. Η κυρία Ρομέρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Ρέντινγκ. Ε, αναγνωρίζουμε το πόσο ικανή είστε στο έργο σας Είχαμε μία Επίτροπο Δικαιοσύνης ε, που πραγματικά έθεσε πάρα πολλά σχέδια, πολλά project επιτάπητος και σας ευχαριστούμε για την ικανότητά σας. Εγώ θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις και σχόλια. Καταρχήν, για πότε έχετε προβλέψει την πρόταση οδηγίας ε, για τη δωρεάν νομική αρρωγή γιατί μιλάμε εδώ για ευπαθείς ομάδες και είναι αλήθεια ότι ε, η ευάλωτη είναι αυτό που ε, μας λείπει, είναι από το πακέτο των οικονομικών δικαιωμάτων και κάποιοι άνθρωποι επειδή ε, δεν έχουν χρήματα δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αν δεν παρουσιάσετε τώρα θα είναι κρίμα γιατί το μόνο που θα λείπει θα είναι η πρόταση για τη δωρεάν νομική συνδρομή. Τώρα ε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία για την ε, πρόσβαση σε δικηγόρο. Ε, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Έχουμε και τη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το άρθρο 6 λέει ότι για μία δίκαιη δίκη ε, πρέπει να παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε ότι έχουμε ολοκληρώσει, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ολοκληρώσει το πακέτο των δικονομικών εγγύσεων όταν μας λείπει αυτό το σημαντικό τμήμα και όταν μιλάμε για το χάρτη πορείας που καταρτίστηκε βάσει του προγράμματος της Οκόλμης ε, συνεχώς αντιμετωπίζαμε δυσκολίες όμως ε, σιγά σιγά ξεπεράσαμε τα τεχνικά προβλήματα όμως εδώ σας παρουσιάζω κάτι που έχει να κάνει με οικονομικούς πόρους γιατί αυτοί που έχουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες είναι οι φτωχοί δηλαδή εμείς τελικά τι κάναμε εκπονήσαμε ένα πακέτο που αφορά μόνο τους πλούσιους γιατί οι φτωχοί δεν έχουν πρόσβαση ε, στη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα ουσιαστικά θέματα και θα έπρεπε να αγωνιστούμε γι' αυτό έτσι ώστε αυτό το πακέτο δικονομικών εγγύσεων να είναι πλήρες. Και δεύτερον, ε, να σας ρωτήσω σχετικά με το σχόλιο που κάνατε για τον Ευρωπαϊκό Αγγελέα και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στο να ορίσουμε το σοβαρό έγκλημα. Δηλαδή, αυτή είναι η βάση που βασίζεται ορισμένε οδηγίε όπω το Eurodac, ε, το PNR. Χρησιμοποιούμε έναν ορισμό που δεν έχει νομική βάση. Εναρμονισμένη. Και με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να θέτει το πρόβλημα. Όταν μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, εμείς ε, ε, πρέπει να αναφερόμαστε στη σύμβαση του παλέρμα γιατί μόνο τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ένα ορισμό καθορίσει. Εμείς δεν έχουμε ευρωπαϊκό ορισμό. Έτσι λοιπόν είναι αδύναμη η βάση αυτών των οδηγίων και θα έπρεπε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προκειμένου να έχουμε κάποιες σταθερές ε, εύρωστες βάσεις και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό που είναι τόσο σημαντικό. Και τέλος για την οδηγία προστασίας των δεδομένων. Ο κανονισμός ε, προχωρά πολύ πιο γρήγορα από την οδηγία, αλλά η οδηγία είναι το πλαίσιο επί του οποίου βασίζονται κατόπιν μια σειρά οδηγιών που κατά κανέναν τρόπο δεν μπορούν να είναι στο περιθώριο αυτής της μεγάλης οδηγίας προστασίας των φυσικών προσώπων. Γιατί τελικά εδώ δεν μιλάμε για προστασία, αλλά για έλλειψη προστασίας των φυσικών προσώπων και σε ορισμένε περιπτώσεις όταν η αστυνομική και η δικαστική συνεργασία το απαιτούν, εμείς ως άτομα δεν είμαστε προστατευμένοι σε σχέση με το πώς ε, είναι αντικειμενικό πώς την χάνουν επεξεργασία στα δικά μας δεδομένα. Θέλουμε να ξέρουμε λοιπόν τις δυσκολίες ε, που υπήρξαν. Γιατί τα τελευταία νέα που είχαμε από την Κυπριακή Προεδρία είναι ότι το Συμβούλιο προτιμά ο κανονισμός να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα και η οδηγία από τη δική μας σκοπιά πρέπει να ακολουθήσει το ρυθμό του κανονισμού γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποιες, ε, κάποια στοιχεία που αφορούν ε, κατασταλτικές πολιτικές ε, στο περιθώριο της προστασίας των δεδομένων, να μην, προστατεύονται λοιπόν τα δεδομένα. Συγγνώμη Πρόεδρε, ένα δευτερόλεπτο μόνο, θέλω να πω κάτι για το έγκλημα στον οικονομικό τομέα αναφερθήκατε στην καταπολέμηση της απάτης και τα λοιπά. Επομένως θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται με τους φορολογικούς παραδείσους. Σίγουρα μπορούμε να μιλήσουμε για πάρα πολλά στοιχεία. Μιλάμε παραδείγματο χάρη για την ασφάλεια των επενδυτών, αλλά δεν μιλάμε για ασφάλεια σε σχέση με τις μεταφορές εισοδημάτων. Και όσο δεν προσεγγίζουμε το θέμα αυτό, δεν μπορούμε να κατολμήσουμε το έγκλημα στον οικονομικό τομέα. Κυρία Ρομέρο, έχουν ζητήσει πάρα πολύ το λόγο και υπάρχουν και άλλοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Έτσι λοιπόν πρέπει πάντοτε να σεβόμαστε το χρόνο, γιατί έχουμε και άλλα σημεία να συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα. Και η κυρία Ρέντινγκ ε, θα πρέπει να έχει και κάποιο χρόνο για να μπορέσει να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που τίθενται. Έτσι λοιπόν σας παρακαλώ να έχετε κατά νου ότι πρέπει να περιορίσετε σε συγκεκριμένα σημεία ή ερωτήματα τα οποία θα απευθύνετε στην κυρία Ρέντινγκ. Η κυρία Φλότρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω πραγματικά ότι για το 2014 αυτό που χρειαζόμαστε για να πείσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες για να θέλουν να ενισχύσουν την Ευρώπη είναι να αποδείξουμε συγκεκριμένα ότι η Ευρώπη ε, χρησιμεύει. Ότι θα έχει ανταποκριθεί στις αιτικές υποχρεώσεις πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και για όλα τα άτομα στην Ευρωπαϊκή Δικαιοδοσία ανεξαρτήτως καταγωγής, φιλετικής, ε, σεξουαλικού προσανατολισμού κλπ και το έχουμε καταφέρει να έχουμε ένωμη τάξη όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Συνδικών θα μπορεί να επιβάλλει στα κράτη-μέλη που μπορεί να υπαναχωρούν λόγω λαϊκισμού, ραζιστικών, ξενοφοβικών κινημάτων να επιβάλλουμε λέγω στα κράτη να σεβόνται τις υποχρεώσεις τους. Και από αυτή την έποψη υπάρχουν δύο θέματα που έθεσαν συνάδελφοι. Είναι το θέμα της στρατηγικής για τη συμπερίληψη των Ρωμά το συζητήσαμε αυτό το θέμα ε, ε, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσω της ένταξης των Ρωμά μπορούμε να αποδείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες διότι είναι τα αντικείμενα ε, διάκρισης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δραστήρια και αποτελεσματική ότι μπορεί να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι όπως κάνατε όταν δεν αυτού αυτούς τους κανόνες στα κράτη-μέλη θα πρέπει να παγιωθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης αυτής της στρατηγικής για την ένταξη των Ρωμά. Σας ρωτώ, τι προβλέψατε σχετικά, πρώτο ερώτημα. Δεύτερο, αυτό που αναφέρθηκε. Εγώ βλέπω ότι θεωρείτε ότι απαντήσετε στην Ολομέλεια όσον αφορά την έκθεση για τη CIA, αλλά δεν ξέρατε ότι αυτή η έκθεση ε, θα τύχανε μεγάλη υποστήριξη. 68 ε, υπέρ, 34 ψήφοι κατά και στην έκθεση γίνονται κάποιες συστάσεις συγκεκριμένες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάναμε πολλέ προσπάθειε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταβάλαμε προσπάθειε το 2007 και φέτο, ούτω ώστε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ανταποκριθούν στι υποχρεώσει του. Μπορείτε, σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υποστηρίξετε, να βοηθήσετε τι χώρε που ακόμα κολυσιεργούν. Και το είδαμε από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, είναι σαφέστατο τώρα. Υπάρχουν ακόμα δύο υποθέσει που εκκρεμωδικούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ρουμανία, Πολωνία, Λιθουανία. Δύο θύματα προσέφυγαν. Α μάθουμε αυτά που συνέβησαν ε, με τη Μακεδονία, λέει ο Μιλήτρια. Ε, τελεσίδικη απόφαση, βασανιστήρια, καταδικάστηκε για τι έκτακτε αυτέ παραδόσει. Μιλάμε και για τι συνέπειε που έχουν αυτά για τα άτομα λόγω τη μεταφορά που έλαβε χώρα από το έδαφο του πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε με θετικό τρόπο αυτό το θέμα εφαρμόζοντας τις συστάσεις, επαναλαμβάνω συγκεκριμένε συστάσεις όπως του πλαισίο ελέγχου και της υποστήριξης εθνικών διαδικασιών όσον αφορά την ανάθεση ευθυνών. Τα κείμενα να μεταφραστούν ούτως ώστε οι έρευνες που ενεργούνται να αλληλοϊποστηρίζονται και θα πρέπει να συντονίσετε τι προσπάθειε που γίνονται στα κράτη-μέλη μέσα των πρωτοβουλίων που δεν να αναλάβετε. Είναι σημαντικότατο λοιπόν για την αξιοπιστία μα. Θα είναι υποφελέ για τι επικείμενε ευρωπαϊκέ εκλογέ του 2014. Η κυρία Χιμένε Θεσσαρίελ, η σειρά σα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την ενεργετική θέση και θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία για να την ευχαριστήσω δημόσια και να τη συγχαρώ για τη δέσμευσή τη να θέσει τα θύματα στη θέση που τους αξίζει και για την αποτελεσματική δεσμευσή της για να τους αποδώσει την αξιοπρέπειά τους. στο πακέτο των θυμάτων ε, που από πρόταση έγινε πραγματικότητα με την έγκριση αυτής της οδηγίας ε, υποστήριξη των δικαιωμάτων και προστασία ε, των θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Να σας πω ότι είναι πάρα πολλοί πολίτες που έρχονται σε επαφή μαζί μου και οι μη καπαόμικρον που πραγματικά σας είναι ευγνώμονες γιατί έχετε βελτιώσει την ασφαλειά τους και τα δικαιώματά τους ε, όταν είναι θύματα σε μια άλλη χώρα πέρα της δική τους. Νομίζω ότι αυτό το νομοθέτημα επαναφέρει την εμπιστοσύνη σε πολλούς πολίτες που σήμερα τη χρειαζόμαστε γιατί υπάρχει μεγάλη δυσπιστία προς τη δικαιοσύνη. Όμως αυτή η οδηγία πρέπει να μετατραπεί σε πραγματικότητα και εγώ σας ζητώ και είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο σας ε, να προβείτε σε παρακολούθηση για το αν διάφορες χώρες εφαρμόζουν αυτή την οδηγία για να μην μείνει νεκρό γράμμα. Όμως εγώ πιστεύω ότι θα το πράξετε και πρόκειται για ένα μέσο που το χρειάζονται οι πολίτες και το ζητούν. Ε, θα ήθελα επίσης να αναγνωρίσω το έργο σας στο ότι προωθείτε την ε, κατάληψη υψηλών θέσεων στις επιχειρήσεις από την πλευρά των γυναικών και θέλω να σα ευχαριστήσω και εκ μέρου τη επιτροπή Γυναικών. Θα ήθελα να σα ρωτήσω, για αυτήν την πρωτοβουλία βρήκατε την απαραίτητη στήριξη, γιατί υπήρχε μεγάλη πολεμική γύρω από αυτό και σε ποιο επίπεδο βρίσκεται σήμερα. Επίση, για να ολοκληρώσω, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, τουλάχιστον οι πολίτες αυτό μας ζητούν και μας ρωτούν, ε, δηλαδή για την ένταξη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να ακούσουμε τα μηνύματα που μας στέλνουν και η ερώτησή μου είναι αν ε, υπάρχουν προτάσεις ε, νομοθετικές ε, που να σχετίζονται με την πρωτοβουλία των πολιτών. Είναι κάτι καλό, αλλά πρέπει να δούμε πώς τα αποτελέσματα θα φτάσουν στους πολίτες και έχετε ουσιαστικά στο νου σας να προχωρήσετε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια πρώτη παρατήρηση. Έχω την εντύπωση ότι ιδιαίτερα σε αυτή την Επιτροπή είναι τόσα πολλά τα θέματα ε, στην ημερήσια διάταξη και τόσο πολυδιάστατα που πάντα έχουμε πρόβλημα χρόνου στη συζήτηση. Και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να συντονίσουμε τις συνεδριάσεις ε, και τα χρονοδιαγράμματα, αλλά μου φαίνεται ότι θα έπρεπε για το θέμα αυτό να αφιερώσουμε μια ολόκληρη απογευματινή συνεδρίαση χωρίς άλλα θέματα για να γίνει σε βάθος συζήτηση όπως πρέπει. Για την έκθεση της κυρίας Ρέντινγκ θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Στις ευρωπαϊκές συνθήκες του Άμστερνταμ, του τα Άμστερνταμ, Νίκια μέχρι Λισαβόνα, πάντα στις συνθήκες είχαμε έναν κανόνα κοινών αξιών και μετά τη Λισαβόνα έχουμε και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ως συστατικό των συνθήκων. Όλα αυτά είναι πολύ καλά. Οι αξίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα, παίζουν ρόλο και είναι καλά. Όμως εγώ έχω την αντίθετη εντύπωση ότι οι αξίες και τα δικαιώματα υπό το πρόσχημα της κρίσης ε, αντιμετωπίζουν μεγάλες πιέσεις και αυτό εγώ το βρίσκω φρεκτό. Το βλέπουμε και στην οδηγία για πρόσβαση σε συνήγορο όπου υπάρχει μια σοβαρή συζήτηση και πολλοί λένε ότι και το δικαίωμα της εμπιστευτικότητας δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, ούτε το δικαίωμα του συνηγόρου, ιδιαίτερα όταν υπάρχει υποψία για τρομοκρατικές πράξεις, ότι πρέπει να κάνουμε εξαίρεση, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου συζητούμε και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι δεν είναι όλοι ύποπτοι για τρομοκρατία τρομοκράτες. Το να πάμε αντίθετα και να πούμε ότι δεν θα πάρεις σε συνήγορο και δεν θα ε, μπορείς να ασκήσεις τα δικαιώματά σου, αυτό το θεωρώ αφόρητο και απαράδεκτο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχω επιφυλάξεις και σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Νομίζω ότι θα είναι υπεύθυνο, πρέπει να είναι υπεύθυνο για, για ένα περιορισμένο τομέα και θα υπάρχει δυνατότητα να επεκταθούν οι αρμοδιότητες. Και ε, όταν είναι ήδη προβληματικό όταν τα δικαιώματα δεν διασφαλίζονται για όλους με τον ίδιο τρόπο. Ένα παράδειγμα, όπου έχω την εντύπωση ότι η κρίση χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τον περιορισμό δικαιωμάτων. Μίλησε για τους διερμηνείς η κυρία Ματιό, που στο Βέλγιο δεν βρέθηκαν λεφτά για διερμηνία. Αυτό πραγματικά είναι πολύ άσχημο, είτε γίνεται στο Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γαλλία ή τη Γερμανία. Είναι πρόσχημα ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά. Εμείς θα πανούμε εκατομμύρια ευρώ για την οδηγία για τα υγρά κλπ. Για τα συστήματα ονομάτων των ε, επιβατών και δε, ξαφνικά δεν μπορεί να πληρωθεί ένας διαρμηνέας και η Ευρωπαϊκή Ένωση όπου τα κράτη-μέλη τώρα ε, ε πάνε να κάνουν περικοπές ε, θέλουν να χρησιμοποιήσουν προσχηματικά λοιπόν τις περικοπές. Επίσης, η οδηγή, ο κανονισμός για την προστασία δεδομένων. Ε, μεγάλα κοντσέρν δραστηριοποιούνται, ομάδες πίεσης και μετά λέμε «Α, οι μικρές επιχειρήσεις επιβαρύνονται τόσο πολύ με αυτά που ζητάμε». Τώρα όμως... Ε, γίνεται μάχη για να εξαιρεθούν ορισμένοι από τις νομοθεσίες μας. Εμείς νομίζω ότι πρέπει ακριβώς να εξετάσουμε καλά τα θεμελιώδη δικαιώματα γιατί όταν δεν έχουν αξία πραγματική τα δικαιώματα και οι αξίες τότε δεν υπάρχει κράτος δικαίου και υπονομεύεται και η δημοκρατία και απειλείται. Ο κύριος Ταβάρες. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ θα προσθέσω κάτι, ίσως υπαθήκαν από τους συναδέλφου Σεντζετίνη, Κύρκοπ, Νταφ, για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ απαιτητική για τα υποψήφια κράτη-μέλη να σέβονται τα κριτήρια της Κοπενχάγης και κατόπιν δεν παρακολουθεί καθόλου τα κριτήρια της Κοπενχάγης αφού έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη. Δηλαδή πώς θα μπορούσε να υπάρχει κάποιο πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς ε, που ουσιαστικά δίνεται κατόπιν τη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά και δεν μπορούν να είναι έτσι τα πράγματα. Ε, Μήπω υπάρχει λοιπόν κάποιο προβληματισμό και κάποιε προτάσει έτσι ώστε να υπάρξει παρακολούθηση για το αν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα τα κράτη-μέλη. Και εγώ θα ήθελα να σας πω ότι θεωρώ ότι η κατάσταση είναι ανεπαρκής. Γιατί, γιατί έχουμε ένα δελτίο ε, όπου επαληθεύουμε την νέα νομοθεσία και να προσπαθούμε ουσιαστικά να κάνουμε τικ ε, σε ε, ότι το χάρη δεν έχει γίνει σεβαστό όμως αυτό δεν αρκεί γιατί ουσιαστικά δεν μπορεί να καλύψει αν υπάρξει γενική αλλαγή της νομοθεσίας έτσι λοιπόν αν υπάρχουν ταυτόχρονα πολλές ε, νομοθετικές αλλαγές, μπορεί να δημιουργηθεί το ακόλουθο φαινόμενο. Καμία από αυτές τις αλλαγές από μόνη της μπορεί να μην παραβιάζει από μόνη της τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά όλες αυτές οι νομοθετικές αλλαγές συλλογικά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ε, ουσιαστικά έλλειψη αξιοπιστίας ε, των δημοκρατικών θεσμών και έτσι λοιπόν μπορεί να έχουμε κίνδυνο να μην γίνονται σεβαστές οι αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της συνθήκης η συστηματική προσέγγιση, να έχουμε αυτό το πίνακα αποτελεσμάτων, ποτέ δεν θα μπορέσει ουσιαστικά να αποτρέψει τις σοβαρότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάτι πιο ποιοτικό και κάτι πιο ερμηνευτικό. Εγώ θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω τι θα πιστεύατε εσείς αν η Ένωση είχε ένα μηχανισμό παρόμοιο με αυτό του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως είναι η Επιτροπή της Βενετίας, δηλαδή πέρα από αυτό το scoreboard, να έχουμε, το χάρη, μία ομάδα εμπειρογνωμόνων που μπορεί να κάνει μία ανάλυση πιο ποιοτική και καθολική για το τι συμβαίνει. Και η Ένωση θα μπορούσε να έχει, το χάρη, μία επιτροπή αντίστοιχη αντίστοιχα τη Κοπενχάγη, να παρακολουθεί αν πληρούνται τα κριτήρια τη Κοπενχάγη στην επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι να μην ε, έχουμε, παραδείγματο χάρη, ε, γενικέ αλλαγέ που τελικά θα δημιουργούν ε, προβλήματα. Ξέρουμε πολλέ φορέ ότι δεν είναι ένα συγκεκριμένο νόμο που θέτει το πρόβλημα, αλλά είναι το αν συμμερίζεται κάποιο ή αν δεν συμμερίζεται και αν σέβεται τι αξίε αυτέ. Και ουσιαστικά ευτυχώς ή δυστυχώς ε, δεν μπορεί να αξιολογηθεί αυτό από το πίνακα αποτελεσμάτων. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η ιδέα, αλλά δεν ξέρω αν θα αρκέσει. Και αν ε, στοιχηματίσουμε μόνο εκεί, ίσως θα δούμε ότι τελικά δεν κάνουμε αυτά που μας ζητούν οι πολίτες, δηλαδή να εγγυηθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως πρέπει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Παπαδοπούλου. Σαν κύριε Πρόεδρε. Απολογούμε γιατί δεν πρόλαβα να ακούσω όλη την ομιλία της κυρίας Ρέτινγκ, αλλά άκουσα τον επίλογο και συμφωνώ απόλυτα για το Ευρωπαϊκό Νέτος Πολιτών. Είμαι και η συγγήτρια. Η πρώτη με ερώτηση επικεντρώνεται για το 2013 Ευρωπαϊκό Νέτος Πολιτών. Επειδή έχει δοθεί μόνο ένας προϋπολογισμός, έναν εκατομμύριο και υπάρχει συζήτηση αν θα γίνει αυτό το ένα, δύο εκατομμύρια ε, διαρωτούμε αν θα είναι αρκετό για να εξασφαλίσουμε εκείνες τις συνέργειες που επιβάλλονται για να πετύχουμε τους δύο στόχους του έτους, που είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η ενημέρωση για τα θεμελιώδη δικαιώματα που απολαμβάνει ο Ευρωπαίος πολίτης λόγω της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας και επίσης η ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε καιρούς οικονομικής κρίσης. Άρα η πρώτη μου ερώτηση είναι για τον προπολογισμό. Και το δεύτερο, θα ήθελα και εγώ να δώσω συνέχεια για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και να ρωτήσω πόσον έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτες και πόσες ε, πρωτοβουλίες, αν γνωρίζετε, έχουν ήδη ε, τροχιοδρομηθεί. Και το δεύτερο ερώτημα μου είναι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχω ακούσει πολλέ εισηγήσει από συναδέλφου, τι οποίε υιοθετώ και υπερθεματίζω. Ε, θεωρώ ότι μιλούμε πολύ και πράττουμε λίγα γιατί ως Κύπρια Ευρωπαία πολίτης βλέπω ότι αυτό το βασικό και πρώτη στο θεμελιώδης δικαίωμα που είναι το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης εργασίας σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζεται σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η δική μου πατρίδα. Και χαίρομαι γιατί ο κύριος Ακυγιάρ έχει πει πολύ έτσι ξεκάθαρα και πολύ όμορφα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυστηρή όσον αφορά τις υποψήφιες χώρες και πρέπει να είναι εξίσου αυστηρή με χώρες μέλη. Εγώ τολμώ να πω ότι δεν είμαστε αυστηροί ούτε για τις χώρες υποένταξη, ούτε με τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εισηγούμε ξεκάθαρα. Ναι, πρέπει να υιοθετήσουμε ένα σύστημα δικτών όσον αφορά το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από υποψήφιες αλλά και από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο, θεωρώ ότι ο κάθε επίτροπος θα πρέπει να δίνει μία ετήσια έκθεση απολογισμού τι έχει κάνει, ποιες πρωτοβουλίες έχει προτείνει, ποιες έχουν υλοποιηθεί, πού βρίσκεται ακριβώς η δράση του και αυτή η έκθεση να μας δίνεται έγκαιρα πριν από το τέλος του χρόνου, να μπορούμε να τη μελετούμε και να ερχόμαστε σε μια συνεδρία στις επιτροπές μας που να έχουμε περισσότερο χρόνο, να μην είναι την τελευταία μέρα που κλείνουμε για τα Χριστούγεννα και να είναι παρόντε όσο το δυνατό περισσότεροι ευρωβουλευτέ για να υπάρχει ένα σωστό και επικοδομητικό διάλογο. Και αυτή η έκθεση να είναι γραπτή και να μα δίνεται τουλάχιστον 10 μέρε πριν για να μπορούμε να τη μελετήσουμε. Τρίτον, θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, το σύστημα, ε, ναι, εκείνο που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνεί οργανισμοί δεν είναι μόνο ψηφίσματα, είναι και μηχανισμοί υλοποίηση. Και τολμώ να πω ότι ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε το Συμβουλίο τη Ευρώπη, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αυτού του μηχανισμού υλοποίηση ψηφισμάτων. Και εδώ χρειάζεται να κάνουμε κάτι πιο δραστικό. Ευχαριστώ. Τώρα είναι η σειρά σας ε, να απαντήσετε κυρία Ρέντινγκ. Ε, είμαι σίγουρος ότι σημειώσατε τα όσα ακούστηκαν. Ε, είχαμε πάρα πολλές σκέψεις και θα σας παρακαλούσα να συνοψίσετε. Θα προσπαθήσω κύριε Πρόεδρε μέσα σε πέντε λεπτά να ανταποκριθώ στο, στα δικαιώματα των βουλευτών και στις ερωτήσεις που κάλυψαν ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο και πολλά θέματα. Πολλές φορές ε, είναι πολύ απαιτητικό και η εργασία μου, γιατί είναι πολύ, πολλά τα θέματα. Το καλύτερο είναι να επικεντρωνόμαστε σε ένα θέμα, ας πούμε, ποινική δικαιοσύνη, αστική δικαιοσύνη, αλλά όταν μιλάμε για τα πάντα και προστασία δεδομένων και θεμελιώδη δικαιώματα και, και, και, δεν είναι δυνατόν να μπούμε στο βάθος όλων των θεμάτων όπως τους αξίζει. Το καταλαβαίνετε νομίζω. Τώρα, αρκετοί από εσάς Ρωτήσατε για την νομική βοήθεια, δωρεάν νομική βοήθεια. Θα θυμάστε ότι αποφάσισα όταν ε, υπέβαλα το σχέδιο οδηγίας ε, για την πρόσβαση σε δικηγόρο, που συνειδητά έβγαλα απ' έξω τη νομική βοήθεια, τη δωρεάν. Γιατί ήξερα ότι αν την είχα προσθέσει, η οδηγία για πρόσβαση σε δικηγόρο δεν θα είχε ποτέ ευοδοθεί. Ήταν πολιτική μου απόφαση που θεώρησα ότι χρειαζόταν τότε για να τα διαχωρίσω αυτά τα δύο. Και σας είπα, ε, ε, επειδή προχώρησαν πολύ τα δικονομικά διαδικαστικά δικαιώματα, ελπίζω ότι θα ολοκληρώσουμε το θέμα της πρόσβασης συνήγορο πολύ σύντομα και μετά θα θέσω επιτάπητο σε ένα πακέτο στο δεύτερο εξάμεινο του 2013 σχετικά με το τεκμήριο αθωότητας, τα ευάλωτα πρόσωπα και τη δωρεάν νομική βοήθεια. Τώρα, κατόπιν τούτου, αν υπάρχει κάποιο στο κοινοβούλιο αυτό που πιστεύει ότι η δωρεάν νομική βοήθεια στα κράτη-μέλη μπορεί να καταβάλλεται μέσα από ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αυτός ο κάποιος κάνει μεγάλο λάθος και δεν χρειάζεται να σας πω σε εσά τους βουλευτές τι γίνεται στις συζητήσεις επί του προϋπολογισμού. Σε όλη αυτή τη διαδικασία μπορούμε να βοηθήσουμε μέσα από την εκπαίδευση κάποιων νομικών. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μαζί με τα κράτη-μέλη, αλλά να πληρώνουμε εμεί την νομική βοήθεια, όχι. Αυτό αποκλείεται. Είναι εκτός των δυνατοτήτων του ε, νοσιακού προϋπολογισμού. Μακάρι να ήταν αλλιώς τα πράγματα, αλλά δεν είναι. Πρέπει λοιπόν αυτά να πληρώνονται από τα κράτη-μέλη λυπάμαι αν η χρηματοδότηση της διερμηνίας που δεν είναι και τόσο μεγάλη, αν ούτε αυτή δεν καλύπτεται. Βέβαια, παντού γίνονται ατυχήματα και ελπίζω να αντιμετωπιστούν μέσα από μέτρα για να μην ξανασυμβούν. Τέτοια πράγματα είναι ατυχή περιστατικά και πρέπει να αποφεύγονται. Διάφοροι συνάδελφοι ρώτησαν για το EPPO, δηλαδή τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, το Ευρωπαϊκό ε, ε, εισαγγελία την Ευρωπαϊκή. Είπα σαφώς ότι θα ε, χαράξουμε το δρόμο προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής εισαγγελία και στο τέλος της εντολής μου θα φροντίσω και θα υποβάλω τη σχετική πρόταση για την δημιουργία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Εμείς αξιοποιήσαμε τις δυνατότητες που είχαμε στην, ε, στο ποινικό δίκαιο, ούτως ώστε να αρχίσουμε με ένα κοινό ορισμό. Για παράδειγμα, τι είναι ένα αδίκημα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Όλα αυτά τα έκανα με τους συναδέλφους μου, που, τους συνεργάτες που είναι υπεύθυνοι για τους φακέλους. Αυτό είναι καθοδόν. Ε, επίσης αρχίσαμε τη διαδικασία μεταρρύθμισης της Eurojust και εδώ προσθέτουμε και το ζήτημα του Γραφείου του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Άρα λοιπόν θα έχετε την πρόταση ε, επιτάπητος για να συνεχίσετε να εργάζεστε σοβαρά όπως ε, είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής σας. Πρόθεσή μου είναι να επικεντρωθώ στην μάχη για την καταπολέμηση ε, αδικημάτων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Ε, είναι το πρώτο βήμα αυτό. Δεν μπορούμε να παραφορτώσουμε τη βάρκα, γιατί αν την φορτώσουμε δεν θα κάνουμε τίποτα. Χρειάζεται προετοιμασία. Τώρα έχουμε τους ορισμούς. Έχουμε τις πρώτες οδηγίες για το ποινικό δίκαιο και όλα αυτά μας πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε θα έρθει φυσικά ε, θα είναι το επόμενο λογικό βήμα στις εργασίες μας. Τώρα, κάνατε αρκετές ερωτήσεις και για τη CIA. Πάρα πολλές φορές έχω έρθει στην Επιτροπή σας για να σας ενημερώσω για τις δυνατότητες που έχει η Κομισιόν να λαμβάνει δράσεις σε αυτό το θέμα και τι έκανε. Έχω δει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, το σημείωσα πάρα πολύ προσεκτικά και απευθύνθηκα με επιστολές στα συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Κάποια από αυτά δεν απάντησαν καν στην επιστολή μου, αλλά είπαν δεν είναι δική σας δουλειά αυτό. Και έχουν δίκιο, γιατί με, τις, βάση τις συνθήκες δεν προβλέπεται να παρεμβαίνουμε εμείς σε τέτοια θέματα. Παρόλα αυτά, παρενέβημεν. Οπότε βλέπετε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει εκείνα να ε, ανταποκριθούν στις ε, υποχρεώσεις τους με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση και με βάση την ομολογία του δικαστηρίου. Γιατί εδώ το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου είναι αρμόδια για τέτοια θέματα. Και εμείς πραγματικά εδώ σε αυτό το θέμα συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ελπίζω κάποια μέρα, όπως προβλέπει και η συνθήκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να, αποτελέσει, να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εμάς, η δική μας η δουλειά ολοκληρώθηκε. Τα περισσότερα κράτη-μέλη θα ήθελαν να προχωρήσουμε στην υπόθεση αυτή, αλλά ένα τουλάχιστον ε, κράτος μέλος, φαντάζεστε ποιο είναι, μας φρενάρει. Ο κύριος Νταφ με ρώτησε για τις εξαιρέσεις που ζητεί το Ηνωμένο Βασίλειο, το opt-out. Έχει αυτή τη δυνατότητα και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και άλλες χώρες μέλη πρέπει να πω. Βέβαια, τη Μεγάλη Βρετανία δεν θα συμμετέχει στο θέμα της πρόσβασης σε δικηγόρο, δεν θα συμμετέχει στο δίκαιο κληρονομίας. Είναι επιζήμιο αυτό για τους Βρετανούς πολίτες, αλλά είναι κυρίαρχη απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης. Τι να κάνουμε. Προβλέπεται από τις συνθήκες το ε, opt-out, οπότε το κάνουν εφόσον θέλουν και αυτό εξαιρούνται. Τώρα, το συνολικό opt-out που έχει ανακοινώσει η Βρετανία, αλλά δεν το πρότεινε συγκεκριμένα μέχρι τώρα, θα εσήμενε ότι θα εξαιρούνταν από 130 νομοθετήματα και κανόνες και μετά θα έπρεπε να ξαναμπούν με διαπραγματεύσεις εξατομικευμένες σε κάθε περίπτωση. Και το είπα Βρετανό Υπουργό Δικαιοσύνης ότι αυτό θα το αναλάβει η επόμενη κυβέρνηση αν το κάνουν και θα είναι πάρα πολύ βλαβερό και για τη δικαιοσύνη και για την ασφάλεια επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν πρέπει να το πολύ συζητάμε, γιατί είναι υποθέσεις αυτές. Εμείς πρέπει να δούμε τα γεγονότα. Τώρα, η μεταρρύθμιση της συνθήκης. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Νταφ ότι καλό θα ήταν να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση νωρίτερα. Και πάντοτε έλεγα ότι θα έπρεπε να το συζητήσουμε αυτό στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας το 2014 και μετά το σχηματισμό της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, το 2014 και να έχουμε και τη σύμβαση το 2015. Όχι ξαφνικά όμως. Και ένας λόγος ε, του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών είναι για να ακούσουμε τους πολίτες, να μας πούν ποιο θέλετε να είναι το μέλλον μας. Θέλετε κι εσείς, όπως εγώ για παράδειγμα, θέλετε να έχουμε ομοσπονδία, να κάνουμε μια ομοσπονδία. Και εγώ το λέω αυτό στο διάλογο με τους πολίτες, το συζητώ, το προβάλλω. Κάποιοι άλλοι θα πούν γιατί δεν το θέλουν αυτό το πράγμα, αλλά θα γίνει συζήτηση και εσείς, όταν θα κατεβείτε στις προεκλογικές σας εκστρατείες, θα βρείτε έτοιμο το έδαφος. Οι πολίτες θα το έχουν ακούσει όλα αυτά. Και θα προβάλλετε κι εσείς το πρόγραμμα που θέλει και το πολιτικό σας κόμμα για το τι πρέπει να γίνει μετά τις εκλογές. Αλλά αυτό πρέπει να είναι ένα σημείο προσυζήτηση στην προεκλογική εκστρατεία. Και γι' αυτό συμφωνώ και με τον κύριο Νταφ ότι όσο νωρίτερα υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προτάσεις της, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Καλό είναι λοιπόν και ευχαριστώ που ασκείτε πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και περισσότερες εξουσίες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό απαντά επίσης σε πολλές ερωτήσεις που ετέθησαν εδώ. Τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Έχετε δίκιο απόλυτο. Έχουμε ένα μέσον για τις χώρες που θέλουν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα μέσο, ένα μηχανισμό για δύο χώρες που ακόμα είναι υπό καθεστώς παρακολούθηση Ρουμανία, Βουλγαρία, αλλά δεν έχουμε μέσον για τα άλλα κράτη-μέλη. Και βλέπουμε ότι δεν πάνε οπωσδήποτε και πολύ καλά τα πράγματα σε κάποια κράτη-μέλη μας. Γι' αυτό ακριβώς υπέβαλα και τώρα έχει ενσωματωθεί μάλιστα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για πρώτη φορά το πίνακα επιδόσεων στη δικαιοσύνη. Είναι θαύμα, συνάδελφοι, που έγινε δεκτός ο πίνακας αυτό το scoreboard στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Τώρα όμως είναι μέσα. Και έχουμε να συσσωρεύουμε τις πρώτες εμπειρίες. Το 2013 θα αναλύεται η λειτουργία των δικαιικών συστημάτων, μάλλον των συστημάτων δικαιοσύνης σε όλα τα κράτη-μέλη, όχι σε όλα, πάνω στη βάση συγκεκριμένων δικτών τους οποίους επεξεργαζόμαστε με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Εκεί κάνουμε κάποια δουλειά πάνω στους δείκτες και αν θέλετε μπορώ να ξαναέρθω κύριε Πρόεδρε και να σας πω λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Πρόκειται για το πρώτο βήμα. Τώρα βάλαμε το πόδι μας στην πόρτα πριν κλείσει και θα υπάρχουν εξελίξεις. Αλλά απογοητεύομαι όταν βλέπω πόσα λίγα μέσα έχω στη διάθεσή μου για την εφαρμογή των κριτηρίων της Κοπενχάγης από τα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που πρέπει να αλλάξουμε σε μια μελλοντική σύμβαση όταν θα αρχίσουμε να συζητούμε για τη μεταρρύθμιση της συνθήκης. Τώρα, το κυβερνοέγκλημα. Αυτά είναι πολύ ξεκάθαρα στο ψηφιακό μας θεματολόγιο. Ε, οι συνάδελφοι Μπαρνιά και Μάλμστρεμ δουλεύουν ε, πολύ εντατικά σε αυτό το θέμα. Ο κύριος Κέρκοπ θα θυμάται ίσως ότι όταν ήμουν Επίτροπος για το ΤΑΚΟΣΕ ήδη είχα διοργανώσει μια διάσκεψη για το κυβερνοέγκλημα και τότε μου είχαν πει τα κράτη-μέλη κάτω τα χέρια. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το λύσουμε εμείς. Πέρασαν χρόνια μέχρι να ξανάρθουμε σε αυτό το θέμα και να καταλάβουμε ότι κανείς δεν μπορεί μόνος του να λύσει αυτό το πρόβλημα. Είναι θέμα που μας απασχολεί όλους και μόνο από κοινού μπορεί να λυθεί. Η κυρία Γιαρόκα, Ζαρόκα, για την οδηγία που ρωτάει. Υπάρχει στην ε, ατζέντα μας το θέμα αυτό. Θα δούμε την ε, εφαρμογή της οδηγίας. Αυτό μοιάζει και με τα θέματα των Ρωμά. Με βάση τα προγράμματα δράσης για τους Ρωμά, μπορέσαμε να δούμε ότι πολλά δικαιώματα είναι στη θεωρία, αλλά όχι στην πράξη. Οπότε κάναμε δύο πράγματα. Πρώτον, είχαμε κάποια σημεία επαφής, κάποιους συνδέσμους στον Ρωμά ε, σε κάθε κράτος μέλος για να μαθαίνουμε τα προβλήματα και έχουμε τώρα μια πιλωτική ομάδα, δημιουργήσαμε μια πιλωτική ομάδα όπου τα κράτη-μέλη, κάποια κράτη-μέλη, εξετάζουν ποια είναι τα προβλήματα που χρειάζονται λύση και για την εκπαίδευση, την υγεία, την εργασία και κάτι άλλο ακόμα. Α, και στέγη, ναι, στέγαση. Σε, αυτό, σε αυτά τα τέσσερα θέματα που υπάρχουν προβλήματα να υπάρξουν λύσεις. Και εγώ θα κινηθώ με βάση τα ευρήματα. Επίσης ασκούνται και πιέσεις από ομολόγους και υπάρχει και σύσταση του Συμβουλίου. Εγώ δεν, τα, δεν το ήθελα αυτό στην αρχή, αλλά τελικά παραδέχτηκα ότι χρειάζεται. Του χρόνου θα υπάρξει ε, σύσταση του Συμβουλίου που δεν θα αντικαταστήσει την ετήσια ανάλυση του τι συνέβη στην πραγματικότητα, αλλά ε, και η πολυπιλωτική ομάδα και οι σύνδεσμοι στα σημεία επαφής που έχουμε για τους Ρώμα ε, θα ε, συμβάλλουν και για το ρατσισμό θα υπάρξει μια έκθεση για την εφαρμογή της απόφασης πλαίσιο και της οδηγίας για την φιλετική ισότητα και αυτά τα δύο θα είναι η βάση, οι δύο εκθέσεις θα είναι η βάση για να αποφασίσουμε αν χρειάζεται περαιτέρω ανάληψη δράσης. Για τα θύματα. Αυτοί οι κανόνες αυξάνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών για το πρόγραμμα δικαιοσύνης μας. Όμως υπάρχει και ένα πρόβλημα. Και ποιο είναι αυτό, ότι οι πολίτες συνήθως δεν είναι ενήμεροι για τα δικαιώματά τους. Και ένας λόγος που υπάρχει το έτος των πολιτών είναι και αυτός. Γιατί το 70% των πολιτών που ρωτήσαμε λένε ότι νιώθουν Ευρωπαίοι, ξέρουν ότι έχουν δικαιώματα και το περίπου 70% πάλι μας λένε ότι δεν ξέρουν όμως ποια είναι τα δικαιώματά τους αυτά. Οπότε δεν είναι αρκετό να ε, προσθέτουμε νέα δικαιώματα. Είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι πολίτες για αυτά τα δικαιώματα, να ξέρουν τι δικαιούνται. Και το γεγονός ότι ε, και να καταλάβουν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαιώματα. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Εκεί έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά ακόμα. Τώρα, η πρωτοβουλία των πολιτών αυτό το χειρίζεται ο κύριο Σεφτσοβιτς. Ε, προχωράει το θέμα, ε, αλλά εδώ είναι σημαντικό όταν συζητήσετε με τον κύριο Σεφτσοβιτς για το πώς προχωρούν τα θέματα να μιλήσετε και για τα προβλήματα και για τα εμπόδια που έχουν οι πολίτες ε, με αυτή την πρωτοβουλία των πολιτών. Τώρα για τις ποσοστώσεις. Τώρα έχουμε μετά από μάχη ένα πρόγραμμα έτοιμο. Ξέρω ότι εδώ στο Κοινοβούλιο θα συνεχίσετε να εργάζεστε πάνω σε αυτό το θέμα. Η συμβολή σας ήταν καθοριστική, γιατί αν δεν είχαν ασκηθεί πιέσεις ε, από το Κοινοβούλιο και από όλες τις πολιτικές ομάδες πρέπει να πω, ε, δεν θα, δεν θα τα είχα βγάλει πέρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Στο Συμβούλιο είναι δύσκολα ακόμα τα πράγματα, αλλά λιγότερο δύσκολα από ό,τι ήταν πριν από λίγους μήνες. Ας πούμε ότι στο Συμβούλιο οι συσχετισμοί είναι ένα τρίτο κατά, ένα τρίτο υπέρ, ένα τρίτο δεν ξέρουν. Οπότε υπάρχει ελπίδα. Ας ασκηθούν πιέσεις στα μέλη του Συμβουλίου που ακόμη δεν έχουν αποφασίσει ή κάποιοι που είναι εναντίον και δεν έχουν διαβάσει το κείμενο. Γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Πολλές φορές μιλάνε ε, θεωρητικά και δεν έχουν διαβάσει πρακτικά το κείμενο. Θα βοηθούσε να διαβάζουν περισσότερο οι πολιτικοί τα κείμενα, τις προτάσεις, ξέρετε. Μάλιστα στο τελευταίο συμβούλιο τους είπα ότι πρέπει να δουν το κείμενο για τις ποσοστώσεις και δεύτερον την ε, συνθήκη και το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Να τα διαβάσουν και αυτό θα βοηθήσει. Καλό είναι κάποιοι υπουργοί να τα μάθουν αυτά τα βασικά κείμενα, να τα γνωρίσουν. Τώρα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και αν αυτά περιορίζονται λόγω της κρίσης. Πολλά πράγματα τώρα περιορίζονται λόγω της κρίσης η κοινωνική ασφάλεια, για παράδειγμα, δεν είναι ε, δικαίωμα θεμελιώδες και όμως αντιμετωπίζει πιέσεις. Ή η φροντίδα των παιδιών, άλλο θεμελιώδες ε, δικαίωμα. Και εδώ υπάρχουν πιέσεις. Οι εθνικοί προϋπολογισμοί ε, περιορίζονται γενικότερα και δυσκολεύουν τα πράγματα όλο και περισσότερο. Γι' αυτό σας λέω ειλικρινά ότι η δωρεάν νομική βοήθεια δεν θα είναι εύκολο πράγμα. Θα δοθεί μάχη για να περάσει από το Συμβούλιο το ζήτημα αυτό, ακριβώς λόγω των πιέσεων στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δεχτούμε. Κάποιο, για κάποιο διάστημα θα έχουμε λιγότερα διαθέσιμα κονδύλια, τα οποία δεν θα μπορούμε να δαπανούμε σε πολύ σημαντικούς τομείς. Παρ' όλα αυτά όμως χρειάζονται όλα αυτά. Για την προστασία των δεδομένων, ε, αυτό το θέλουμε, ακόμα και αν ασκούνται πιέσεις. Βλέπω εδώ τον κύριο Άλμπρεχτ. Ρωτήστε τον για το lobbying. Βλέπω και τον κύριο Δρούτσα εκεί. Ρωτήστε τους για το lobbying. Πολλοί ξέρετε ότι η άσκηση πιέσεων άρχισε και πριν υποβληθεί το κείμενο. Ε, οι lobbyists προσπάθησαν να με πιέσουν για να ε, άσκησαν πιέσει σε σχέση με το κείμενο. Υπάρχει το κείμενο παρά το lobbying και έχετε ένα ολόκληρο πακέτο. Κανονισμό και οδηγία. Εγώ επιμένω στο πακέτο. Οι συγητές επιμένουν στο πακέτο. Και δεν αφήνουμε κανέναν να υποσκάψει το πακέτο και να το ανατρέψει. Ήταν, είναι, θα έλουμε να είναι πακέτο. Και δεν θα κάνουμε αναγκαστικά αυτό που μας λέει η μία ή η άλλη Προεδρία. Τελεία και παύλα. Η Ιρλανδική Προεδρία έθεσε την προστασία δεδομένων ως ε, μία βασική προτεραιότητα και εμείς το καλωσορίζουμε αυτό, παρόλο που είναι δύσκολο. Και θα ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση που έδωσε η Προεδρία εκείνη. Το έτος του πολίτη έχει προϋπολογισμό ένα εκατομμύριο μόνο. Μάλιστα. Μακάρι να είχε περισσότερα. Αλλά θα το δουλέψουμε ακόμα και έτσι, χωρίς παραπάνω λεφτά αρχίσαμε παντού και με τη βοήθεια των, ε, ευρωβουλευτών, των βουλευτών στις ε, περιοχές. Ε, είχαμε τις πρώτες συνεδριάσεις των δημαρχείων. Πρέπει να σας πω ότι χαίρονται που επιτέλους έρχεται κάποιος να τους βρει, να καθίσει κάτω και να τους ακούσει. Σας λέω την εμπειρία μου από τις τρεις μεγάλες ε, συναντήσεις ε, σε δημαρχιακό επίπεδο. Ε, ο, ο κόσμος δεν είναι επιθετικός, είναι ευγνώμων που έρχονται οι πολιτικοί σε εκείνο το επίπεδο για να, να συζητήσουν και να ακούσουν. Δεύτερον, ε, υπάρχουν πολλά αιτήματα για περισσότερη Ευρώπη. Και όταν τους εξηγώ ότι αυτό εγώ δεν μπορώ να το κάνω γιατί δεν προβλέπεται από τη συνθήκη, μου λένε τότε, ε τότε άλλαξε τη συνθήκη. <laughs> Εύκολο βέβαια το λένε αυτό οι πολίτες βέβαια. Λύστε το πρόβλημα. Δεν ξέρουν τις δυσκολίες της δημιουργίας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, δεν ξέρουν πόσο περίπλοκο είναι να συνταχθεί νέα συνθήκη, αλλά τα αιτήματά τους είναι πολλά ε, προς εμάς. Και βέβαια ε, όλα αυτά θα παίξουν μεγάλο ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία. Γιατί τότε πρέπει να ξέρουμε τι ζητάνε από εμά οι πολίτες και πώς θα αντιδράσουμε εμείς του χρόνου κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών και βέβαια και τι θα κάνουν και τα πολιτικά κόμματα που θα κατέβουν στην προεκλογική μάχη. Για την ελεύθερη διακίνηση μία πληροφορία θα σας δώσω. Όταν ανέλησα την οδηγία για την ελεύθερη διακίνηση, γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα με τη Γαλλία, θα θυμάστε, ήταν το ζήτημα των Ρωμά. Ε, πρόσεξα ότι 16 κράτη-μέλη δεν είχαν εφαρμόσει σωστά την οδηγία για την ελεύθερη διακίνηση. 10 από αυτά το έκαναν τώρα, τα 6 τα πήγα στο δικαστήριο. Ευχαριστούμε κύριε Ρέντινγκ. Ε, Διέρχεστε σχεδόν δύο ώρες τη συζήτηση αυτή και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να παραπονεθεί σε αυτή τη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΠΕ για το πόσο ευέλικτα διαχειριζόμαστε το χρόνο, γιατί βάζουμε τα δυνατά μας. Όχι μόνο ε, να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά να μπορέσουμε να ακούσουμε και όλες τις ιδέες που πρέπει να ακούσουμε με τη συζήτηση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ρέντινγκ που ήταν εδώ μέχρι τελευταία στιγμή. και σας ευχαριστούμε που απαντήσετε τόσο προσεκτικά σε κάθε μεμονωμένη ερώτηση και δείξατε την πότητα να συνεχίσετε τη συνεργασία ενεργετικά. Ανυπομονούμε να ε, συνεχίσουμε τη συνεργασία και εγώ ως εισηγητής για αυτήν την ενδιάμεση αναθεώρηση του πρόγραμματος της Οκόλμης. Ε, σας ευχόμαστε να είστε καλά και καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά.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 λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο αλλά και την σημερινή ημερομηνία γιατί είναι η τελευταία μέρα εργασία για πολλού από εμά εδώ, όχι για όλου, αλλά για ορισμένου εξήμων τουλάχιστον. Αυτή είναι η τελευταία τακτική συνεδρίαση τη Επιτροπή μα ε, πριν από τι χριστουγεννιάτικε διακοπέ. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Πρίμπε που βρίσκεται εδώ. Τον κύριο Ράινφερτ Πρίμπε που βρίσκεται εδώ. και τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την παρουσίασή του για την ε, δεύτερη κοινή επεξέταση τη εφαρμογή τη συμφωνία TFTP, του προγράμματο παρακολούθηση χρηματοδότηση τρομοκρατία που μόλι δημοσιεύθηκε από την Κομισιόν 14 Δεκεμβρίου και κυκλοφόρησε, διανεμήθηκε σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Για τα επόμενα 10 λεπτά θα ακούσουμε την παρουσίαση του κ. Πρίμπε και κατόπιν θα ανοίξουμε τη συζήτηση. Να σας πω τώρα το επόμενο σημείο, το σημείο 14, που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου περί του καταλόγου τριτών χωρών, υπήκοοι των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση θεώρηση για τη διέλευση των εξωτερικών σανόρων των κρατών μελών και του καταλόγου των τριών χωρών υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Αρμόδιος συζητής είναι ο κύριος ε, Αγουστίνη Δίας Δεμέρα δεν ε, θα λάβει χώρα, αναβάλλεται. Γιατί ο κύριος Μέρα δεν μπορεί να τα καταφέρει σήμερα να παραβρεθεί εδώ. Επομένως, περνάμε στο επόμενο σημείο, που θα περάσουμε μάλλον στο επόμενο σημείο, που θα είναι το σημείο 18. Και αν τα καταφέρουμε να κινηθούμε γρήγορα, μάλλον θα κάνουμε παράκαμψη θα ολοκληρώσουμε πριν από την ορισμένη ώρα της συνεδρία μας. Λοιπόν, έχετε το λόγο κύριε Πρίμπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε και καλό απόγευμα σε όλους. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την έκθεση για την δεύτερη επανεξέταση της ε, συμφωνίας εφαρμογής ε, Συμφωνία τη FTP μεταξύ ΕΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Στι αρχέ του περασμένου έτου κάναμε την πρώτη αξιολόγηση και βάσει δύο συναντήσεων που είχαμε. Αυτή τη φορά είχαμε μια συνάντηση στη Χάγη για να εξετάσουμε την ειδική συμμετοχή της Europol και η δεύτερη συνεδρίαση έλαβε χώρα 30 και 31 Οκτωβρίου στην Ουόσικτον. Και εκεί είχαμε και τον τυφώνα Σάντι, όπως γνωρίζετε τότε, και ολοκληρώσαμε την έκθεση αυτή την περασμένη εβδομάδα. Είναι αποτέλεσμα εντατικού διαλόγου με τις Αμερικανικές Αρχές και πρέπει να πούμε ότι εκτιμούμε πως από την Αμερικανική πλευρά και πάλι αυτή η αναθεώρηση προετοιμάστηκε πάρα πολύ καλά και μας επέτρεψε να συζητήσουμε όλα τα θέματα που θέλαμε να συζητήσουμε μαζί τους. Όπως θα είδατε πιθανότατα στην έκθεση, η ε, Πάνεξέταση του προγράμματος παρακολούθησης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για την καταπολέμηση και την πρόληψη της τρομοκρατίας. Ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η συνεχίζει να ωφελεί την Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτές τις αμοιβέ διευθετήσεις ε, και όπως θα δείτε αναφέρουμε και το θέμα της αμοιβαιότητας στην έκθεσή μας. Ε, ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό παράδειγμα που εξετάστηκε είναι η περίπτωση όπου κάποιες πληροφορίες βοήθησαν τη Γεροπόλη και άλλους Ευρωπαίους ερευνητές αλλά και ερευνητές να ε, βρουν ε, ουσιαστικά ε, πώς είχε γίνει η χρηματοδότηση για κάποιες τρομοκρατικές επιθέσεις. Και επίσης οι αρχές ενός κράτους μέλους σε άλλη υπόθεση μπορούσαν να συλλάβουν ένα άτομο ο οποίος είχε σκοπό να χτυπήσει πολιτικούς στόχους. Και ε, ε, ακολουθούμε ασφαλιστικέ ασφαλιστικές οι συστάσεις που παρουσιάστηκαν στην πρώτη έκθεση το Μάρτιο του 2011 σε μεγάλο βαθμό ακολουθήθηκαν και το ελέγξαμε αυτό, ε, αφιερώσαμε τον κατάλληλο χρώμα και έτσι βελτιώθηκε η εφαρμογή τη συμφωνία. Βέβαια, Σημαντικέ περαιτέρω βελτιώσει έλαβαν χώρα, κυρίω σε ό,τι αφορά τι λειτουργίε επαλήθευση και εποπτεία που πάνε πέρα από όσο απαιτεί η συμφωνία. Η συνεχιζόμενη διαδικασία διαδικασία της διαγραφής δεδομένων παλιότερων των πέντε ετών είναι ένα ζήτημα που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση γιατί εδώ εντοπίσαμε κάποια ελλείμματα που αναγνωρίστηκαν από τις Αμερικανικές αρχές. Και έχουμε την ευκαιρία στην κοινή έκθεση αναξιολόγησης ε, ε, να το ξαναδούμε αυτό στα μέσα του 2013, όπως ε, απαιτείται από την συμφωνία. Για να πω τώρα σε κάποιες λεπτομέρειες, χωρίς να διαβάσω και πάλι όλη την έκθεση, θα δείτε στην έκθεση. Ξεκινάμε με τη σελίδα 4. Εκεί αναφερθήκαμε στα στατιστικά στοιχεία που έχουμε και κατανοούμε με σαφήνεια τη διάσταση της χρήσης των δεδομένων, κυρίως ό,τι αφορά τις έρευνες. Υπήρξε μείωση του αριθμού των έρευνων που μπορεί να χρειάζονταν και καλύπτονταν από την πρώτη έκθεση. Υπήρξε κάποια καθυστέρηση, κάποιο φόρτο εργασίας, επειδή δεν υπήρξαν διευθετήσεις πριν να τεθεί σε συμφωνία. Επίσης, εξετάσαμε εις βάθος τη λειτουργία του μηχανισμού του άρθρου 4, δηλαδή την επαλήθευση του αιτήματο από το Υπουργείο Οικονομικών, από το SWIFT και όπως βλέπετε στην έκθεση υπήρξαν σαφείς ε, βελτιώσεις εδώ λόγω διαφορών παραγόντων. Καταρχήν, ε, η ίδια η Europol είχε φέρει αντίρρηση σε κάποια από τα αιτήματα στο αρχικό στάδιο της συμφωνίας, αλλά, και επίση να το πούμε και πολύ σαφώς, η όθηση που δόθηκε από την JSP της Europol. Επίσης, έπρεπε να διερευνήσει τις δυνατότητες να καταστήσει πιο στιασμένες ε, τις αιτιάσεις των ΗΠΑ. Και υπήρξε εκεί η δυνατότητα να δει κάποιες απόρριτες αιτήσει και να συγκρίνει τις αιτήσει που είχαν γίνει στους πρώτους μήνες της συμφωνίας με κάποιες μετέπειτα ε, αιτήσει και τη διεκπαιρέωσή του τώρα. Και όλα τα μέλη της ομάδας διέγνωσαν σημαντική πρόοδο και αυτό σημαίνει και το βλέπετε αυτό στο κουτί των συστάσεων. Η σύστασή μας είναι να συνεχιστεί αυτή η επαλήθευση υψηλών προτύπων. Αυτά είναι καλά νέα λοιπόν. Επίσης, ε, είχαμε ένα νέο μηχανισμό, είχαμε ένα phasing in, να έχουμε εποπτεία από ένα δημόσιο φορέα για να εξετάζει πώς ε, γίνονται οι έρευνες. Και πριν ε, από χρόνια ε, είχε ζητηθεί αυτό από μία συναδελφό σας. Έτσι λοιπόν τώρα προετοιμάζουμε μία δεύτερη εκδοχή αυτού του μηχανισμού και κάτι που είναι σημαντικό και το τονίσαμε στην έκθεση είναι ότι υπάρχει μια ομαλή συμπληρωματικότητα μεταξύ της εταιρείας ε, ε, και της Κομισιόν γιατί γίνεται επιμερισμό της εργασίας. Έτσι λοιπόν αυτή η συνεργασία μεταξύ των εποπτών τώρα λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Τώρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων και τα δικαιώματα που συνδέονται ε, με την προστασία των δεδομένων, δηλαδή και όμως πρόσβαση στα δεδομένα, διόρθωσης κτλ. Μα εντυπωσίασε το ότι υπάρχουν πάρα πολύ λίγα αιτήματα από τους πολίτες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. έχουμε αυτή την ε, γραμμή επικοινωνίας ε, για τις επιχειρήσεις ε, γιατί, όταν, βλέπουμε εκεί ότι ενδιαφέρθηκαν πάρα περισσότερο για τις κυρώσεις που μπορεί να επιβάλλονται στο Ιράν παρά για την συμφωνία τη FTP και τα σχετικά δεδομένα. Κατόπιν στη σελίδα 12 της έκθεσης θα δείτε κάτι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Έχουμε κάποιες διατάξεις που έχουν να κάνουν με την αμοιβαιότητα, σε ποιο βαθμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ποια είναι η ασφάλεια, με στην Ευρωπαϊκή Ένωση πόσο ωφελούμαστε από τα δεδομένα TFTP. Εδώ σημειώσαμε ότι υπάρχει εξέλιξη. Ζητούμε από τα κράτη-μέλη άρθρο 10 βάσει του άρθρου 10 ε, αυξάνονται οι αιτήσει, όμως ε, εκεί είχαμε κάποια δυσκολία διερεύνησης, γιατί σύμφωνα με τη συμφωνία αυτά τα αιτήματα στέλνονται μέσω της Europol ή απευθείας στέλνονται από τις αρχές των κρατών μελών. Και αυτές οι αρχές των κρατών μελών θα μπορούσαν να είναι είτε διοκτικές αστυνομικές αρχές δηλαδή, είτε μυστικές υπηρεσίες. Και ρωτήσαμε τα κρατημέλη σχετικά με τα θέματα αυτά και βλέπετε κάποιες ενδείξεις, αλλά μπορεί να υπάρχουν κάποια ελληματικά στοιχεία εκεί. Γιατί τα κρατημέλη μπορεί να μην ήταν έτοιμα να μας δώσουν ακριβείς πληροφορίες και βλέπετε στις συστάσεις ε, ότι έχουμε αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό. Και ζητώ συγγνώμη που θα επανέλθω σε ένα θέμα προστασίας των δεδομένων, το οποίο το παρέλειψα. Τη διαγραφή των δεδομένων γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τη συμφωνία φέτος τον Ιούλιο τα δεδομένα παλιότερα των πεντετών έπρεπε να διαγραφούν. Αυτό έγινε. Και μας εξήγησαν οι Αμερικανικές Αρχές λεπτομερώς ότι για τεχνικούς λόγους τέτοια διαγραφή δεν μπορεί να γίνεται κάθε μέρα. Πρέπει να γίνεται σε κάποιες συγκεκριμένες καθορισμένες περιόδους. Δεν είναι δηλαδή εύκολο να διαχωριστούν τα παλιά από τα νέα δεδομένα. και συνειδητοποιήσαμε ότι ο τρόπος που το κάνουν τώρα δεν είναι και απόλυτα ορθό. Γιατί η αρχική πρόθεση ήταν ε, να τα διαγράψουν τον επόμενο χρόνο τον Ιούλιο. Και αυτό θα σημαίνει ότι θα υπήρχαν κάποια δεδομένα που θα ξεπερνούσαν τα πέντε έτη κατά κάποιους μήνε στην παλαιότητά τους. Όμως ε, βλέπετε εδώ ότι αυτά ε, μας τα είπαν μετά την ε, επισκόπηση και έτσι λοιπόν η επισκόπηση έχει άμεσα αποτελέσματα για την αλλαγή του συστήματος γιατί παρακολουθούμε στενά αυτό το ζήτημα. Και το σημείο 217 σελίδα 14 εδώ η έκθεση δηλώνει με σαφήνεια πόσο σημαντικό θεωρείται αυτό το μέσο από τις Αμερικανικές Αρχές. Δεν θα σας κλείσει αυτό βέβαια. Αλλά και για τη δική μας ε, ασφάλεια και από τι δικέ μα ε, αρχές ε, θεωρείται σημαντικό. Είχαμε μια συζήτηση για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τη διαφάνεια αυτού του μηχανισμού. και οι αμερικανικέ αρχές ανησυχούν ε, να μην διακινδυνεύσουν το απόρριτο μιας επιχείρησης. Όμως λέγεται σαφώ την έκθεση ότι πρέπει να γίνουν κάποιες περαιτέρω προσπάθειες. Να είμαστε κάπω πιο ανοιχτοί και να εξηγούμε πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός ε, και ποια είναι η προσθεμένη αξία. Και τέλος, σελίδα 15 και σελίδα 16 βλέπετε κάποιες σκέψεις ε, για τη διαδικασία της αναθεώρησης. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η διαδικασία επανεξέτασης ε, και συνειδητοποίησαμε ότι είναι μια συνεχής διαδικασία. Δηλαδή δεν έχουμε ένα ραντεβού μόνο κάθε 18 μήνες, αλλά σε όλα τα επίπεδα, σε επίπεδο κομισιών, ε, επίπεδο ε, τεχνικό, όλα τα επίπεδα αξιολογήθηκαν και προσπαθήσαμε να βρούμε τις διάφορες δυσκολίες. Ίσως υπήρχε κάποια σύγχυση για το πώς ε, η διαδικασία επαναξέτασης θα πρέπει να συνδέεται και με άλλες πρωτοβουλίες. Και η Κομισιόν μας ζητά να κάνουμε όσα λέει συμφωνία, δηλαδή να διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζεται σωστά ο μηχανισμός αυτός μέσω της διαδικασίας επανεξέτασης. Και θα βρείτε κάποιες συστάσεις στη σελίδα 16 σχετικά με το ζήτημα αυτό. Όλες οι συστάσεις συνοψίζονται στο τέλος της έκθεσης και θα ήθελα να κλείσω ευθύντας την προσοχή σας στα παραρτήματα για την, ε, όπως και για την τελευταία έκθεση, είχαμε ένα μακροσκελές παράρτημα 1, όπου δίνονται οι λεπτομερείς απαντήσεις των Αμερικανικών αρχών για ένα σύνολο 42 θεμάτων, ερωτήσεων που συζητήσαμε μαζί τους και συζητήσαμε το σχέδιο των απαντήσεων στη συνάντηση στην Ουάσιγκτον. Θα μπορούσε κάποιο να πει ότι αυτό το τμήμα, σελίδα 19 έως και 34, είναι ίσως και πιο σημαντικό από την κυρία έκθεση. Γιατί εκεί περιλαμβάνονται πάρα πολλές λεπτομερείς πληροφορίες. Και θα πρέπει να ειδωθεί ως ένα συμπληρωματικό τμήμα της έκθεσης. Θα δείτε και στο παράρτημα 3 τα στατιστικά στοιχεία που σας ανέφερα για το πώς λειτουργεί η Europol και νομίζω ότι κάποια μέλη αυτής της Επιτροπής ε, ζήτησαν κάτι συγκεκριμένο. Συζητήσαμε ορισμένες υποθέσεις ε, όπου έχουμε παραδείγματα για το πώς χρησιμοποιήθηκε η TFTP και θεωρήθηκε χρήσιμη από τις Αμερικανικές αρχές. Τώρα, ο δρόμος προς τα μπρος. Έχουμε δύο ραντεβού για μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 της Συμφωνίας. Η Κομισιόν ε, και το Υπουργείο Οικονομικών θα παρουσιάσουν μια κοινή έκθεση σε ό,τι αφορά την αξία της TFTP, δίνοντας στοιχεία το εργότερο μέσα σε τρία χρόνια από τη θέση σε ίσχυ της συμφωνίας. Δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο του χρόνου θα έχουμε αυτή την κοινή έκθεση και μέχρι την ίδια ημερομηνία η Κομισιόν θα παρουσιάσει μία έκθεση προόδου για την εξέλιξη ενός ισοδύναμου συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά το άρθρο 11 της Συμφωνίας, όπως κληθήκαμε ε, στην απόφαση του Συμβουλίου που ενέκρινε τη συμφωνία αυτή. Και πρόσθετα συμφωνήσαμε με τις Αμερικανικές Αρχές ότι η επόμενη κοινή επαναξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 13, θα υλοποιηθεί το 2014. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσει η συζήτηση. Ξεκινάμε από τη Σοφή Ιντβελτ, την Αντιπρόεδρο. Θε να πάει στο λόγο, Σοφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρίμπε που βρήκατε χρόνο για να μας ενημερώσετε σε αυτό το περίπλοκο θέμα εδώ στο Κοινοβούλιο. Μας απασχολεί τόσο καιρό. Νομίζω ότι ε, έχετε κάνει πολλά στα πλαίσια της ιδέας της Κομισιόν. Τώρα, καλό θα ήταν να δούμε πιο συγκεκριμένα Πού υπάρχουν ελλείμματα εκτός από αυτά που μας είπατε ε, για τις περιόδους διαγραφής ε, των δεδομένων ότι γίνεται σχεδόν σε αιτήσια βάση και όχι κάθε πέντε χρόνια. Χωρίς ε, να θέλω να κάνω κακοπροαίρετες ερμηνείες, νομίζω ότι πολλά θέματα έχουν παραμείνει ανοιχτά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, αλλά θέλω να αναφέρω ορισμένα προφανή. Σε σχέση με το άρθρο 4, την εντολή, τα δεδομένα να έχουν συγκεκριμένη μορφή όταν διαβιβάζονται ε, και υπάρχει η οδηγία ένα μεγάλο κομμάτι, αν όχι το μεγαλύτερο, να Πολλά δεν δίνονται με τη μορφή που πρέπει, αλλά ε, παραμένουν, ε, ε, έχουν όλα διαβιβαστεί στη ΣΥΠΑ και παραμένουν σε μια μορφή όπου μένουν εκεί χωρίς να γίνεται πολύ χρήση των στοιχείων αυτών. Στην έκθεση παρουσιάζονται οι ε, πώς αναζητούν, οι αναζητήσεις, ε, αλλά όχι πόσες, ε, πόσα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι δεν υπάρχουν αναζητήσεις Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό δεν εκπλήσει γιατί προβλέπεται να περνούν μέσω του εθνικού εντεταλμένου. Γι' αυτό δεν φτάνουν μέχρι το Υπουργείο Οικονομικών. Όμως ε, δημιουργήθηκε ένα δικαίωμα και το είπε η κυρία Ρέντινγκ πριν και όταν δημιουργούνται δικαιώματα θα πρέπει αυτά να μπορούν να εξασκούνται. Είναι, όπως ε, είπατε και την προηγούμενη φορά, είναι δύσκολο να μάθουμε αν τα δεδομένα με τις δικές μου χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, που μπορεί να μην είναι ενδιαφέρουσες αλλά γίνονται, εάν ε, υπάρχουν δεδομένα για αυτές. Είχαμε κάνει συναντήσεις ε, με τον ε, ε, υπεύθυνο και μάθαμε ότι υπάρχουν δεδομένα που διαβιβάζονται ακόμα και στοιχεία σχετικά με το δίπλωμα οδήγησης. Και μετά από δύο χρόνια δεν έχουμε στοιχεία σχετικά με τα δεδομένα αυτά, εκτός και αν Ναι, υπάρχει τεχνικό πρόβλημα γιατί το μέχρι πριν από... Έκλεισαν όλα τα μικρόφωνα, ο πρόεδρος είναι χωρίς μικρόφωνο. Αλλά όταν ομιλούσε ο κύριος Άλβαρ ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο του πρόεδρου και είχαμε πρόβλημα για να ακούσουμε. Ναι, τώρα έκλεισε το μικρόφωνο. Ο πρόεδρος λέει ότι δεν έχει ανοιχτό μικρόφωνο στο Προεδρείο, αλλά είχε. όχι, κινητό δεν είχα. Αν είχα κινητό, λέει ο κύριο Άλβαρο, θα ενοχλούσε. Εν πάση περιπτώσει, αν, έχω, αν υπάρχει θόρυβος, πείτε μου, αν δεν την ακούτε, λέει ο κύριο Άλβαρο. Λοιπόν, τέλος. Τρία σημεία ακόμα θέλω να αναφέρω. Το θέμα της αναγκαιότητας και της αποτελεσματικότητας. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Μπορούμε να πούμε ότι είναι θέμα συσταλτικής ή διασταλτικής ερμηνείας της αναλογικότητας. Υπάρχουν 57 leads μέχρι τώρα μέσα σε δύο μήνες περίπου, ένα ε, για κάθε κράτος μέλος το χρόνο. Επίσης, θα πούν και οι συνάδελφοι και άλλα θέματα, εγώ περιορίζομαι σε δύο. Πρώτον, χάρηκα που είπατε ότι τον Αύγουστο όταν θα έρθει η οριστική έκθεση θα δούμε ε, για το σύστημα, το σύστημα των εκδόσεων και τη διαδικασία. Ε, επίσης αυτό που είπε η Επίτροπος με ενδιαφέρει σχετικά με το ότι δεν συνεχίζουμε τις εναλλακτικές που ήταν τρεις νομίζω σε μια ανακοίνωση που δόθηκε. Αυτό όμως ήταν βασική προϋπόθεση γιατί ε, συμφώνησαν με τη διαδικασία αυτή ε, πολλοί βουλευτές και με αυτή την συμφωνία. Ήταν σημαντικό ε, ότι δόθηκαν προσωπικές διασφαλίσεις σε βουλευτές δεν μπορεί δηλαδή να τα βλέπουμε αυτά επιπόλαια, τα υπεσχημένα πρέπει να τηρούνται. Επίσης ε, είπε η Επίτροπος ότι δεν υπάρχει ε, πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Υπάρχει όμως ε, για την νομοθεσία και το άλλο, η άλλη αρχή που είναι αρμόδια, το Κοινοβούλιο. Και Νομίζω ότι αν δεν ε, ενημερωνόμαστε κι εμείς ε, ε, και δεν συμφωνούμε δεν μπορεί να λειτουργήσει η νομοθεσία. Τέλος, η συμφωνία αυτή δεν μπορεί στο μέλλον να μην, τη τη χρειαζόμαστε με αυτή τη μορφή και βέβαια περιμένω να δω τι θα γίνει μετά τον Αύγουστο. Εγώ καλώ και τις, και τις έχω καλέσει και επανειλημμένα τις άλλες ομάδες να συνεργαστούν μαζί μου και να σκεφτούμε αν δεν υπάρχει ε, εκπλήρωση των υποχρεώσεων, να δούμε μήπως μπορούμε να αναστείλουμε την ε, διαδικασία. Μπορεί δηλαδή εμείς να είμαστε σε θέση να απαντούμε εξατομικευμένα στα αιτήματα των Αμερικανών, να τους δίνουμε τα στοιχεία που θέλουν, όχι όμως να διαιωνίσουμε ένα σύστημα μαζικής διαβίβασης δεδομένων επ' αυτής της βάσεως ε, έγινε συμφωνία με το Κοινοβούλιο και συμφώνησε το Κοινοβούλιο και αυτό πρέπει να το τηρήσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ματιού έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είχαμε την έξοδο 2011 και τώρα έχουμε αυτή μπροστά μας. Συνέβησαν πρόοδοι στη Μεσοπερίδιοδο. Η σύσταση του 2011, η συστάση του 2011 απεφαρμόστηκαν εθέρω τη διαδικασία εφαρμογή συμφωνία και εφαρμογή του, η θέσπιση του υπευθύνου για τα δεδομένα, Πριν να τα σημειώσουμε. Κατανοώ αυτά που είπατε κύριε Αλβάρο, αληθεύουν, αλλά θα πρέπει να πούμε και όλα αυτά που συνέβησαν μεταξύ της εκθέσεως του 2011 και τώρα. Έχουμε και την Ευρωπόλη η οποία σημείωσε πρόοδο. Ε, λοιπόν, εφάρμοσε τις διάφορες συστάσεις Ευρωπόλ, επικοινωνούσε με την ε, αρμόδια αρχή μέσω διοργανώσεως κοινών ομάδων εργασίας. Κάτι που μας ικανοποιεί. Καλή δουλειά της Ευρωπόλ. Βελτίωσε τη διαδικασία της επαλήθευσης. Βελτίωσε τη διαφάνεια. Βελτίωσε τη συνεργασία με, τις, με την κοινή αρχή. Σημαντικό. Εμείς διορίσαμε την ευρωπόλη για τη εβίβαση των στοιχείων. Είναι μια συμφωνία δύσκολο να εφαρμοστεί. Το Κοινοβούλιο ήθελε να την εφαρμόσει. Ακόμα και αν δεν είναι αιώνια πρέπει να, ε, να λειτουργήσει μέχρι την εκπνοή της. Μας εξυπηρέτησε εν γέννη, ο κ. Πριμπέ αναφέρθηκε σε κάποια παράδειγματα που για του Ολυμπιακού Αγώνε του Λονδίνου. Ήταν πολύ χρήσιμη και πρέπει να το πούμε και σε άλλε περιστάσει. Η ασφάλεια των πολιτών, μην το λησμονούμε, είναι θεμελιώδε δικαίωμα. Το υπενθυμίζω. Και αυτή η συμφωνία σημαντικότατη. Πολύ συχνά τα κράτη-μέλη καλούν τη ΣΥΠΑ για την αποστολή πληροφοριών. Πρέπει να το έχουμε υπόψη και αυτό. Θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια διαδικασίε. Πιο ασφαλεί διαδικασίε. Όμως Πρέπει να ωφεληθούμε όσο δυνατόν περισσότερο χρόνο από αυτή τη συμφωνία κατά την απόψή μου. Είναι μια συμφωνία που για την ώρα ακόμα και αν μπορεί να είναι καλύτερη όσον αφορά κάποιε διαδικασίε, αν θα μπορούσε να βελτιωθεί, όσον αφορά τι διαδικασίε, πιστεύω ότι αν δεν την παρατείνουμε, ε, δεν θα είναι καλό. Σκεφτείτε πόσα ωφέλη έδωσε στην καταπολέμηση τη τρομοκρατία και πόσο υποφελέ είναι αυτό για τον Ευρωπαίο πολίτη, για του Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ, η κυρία Τσίμπελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια θεμελιώδης εισαγωγική παρατήρηση. Είναι σημαντικό κοινοβούλιο ευρωπαϊκό κάποια στιγμή να έχουμε μια ρύθμιση, να βρούμε μια ρύθμιση για να βλέπουμε απόρριτα κείμενα. Δεν είναι δυνατόν να θεωρούνται απόρριτα κάποια κείμενα, να μην μπορούμε να τα δούμε εμείς και γι' αυτό να μας λείπουν πληροφορίες για να μπορέσουμε να κρίνουμε πού είναι το πρόβλημα. Και βέβαια στο μέλλον δεν θέλω να βάλω στον πειρασμό καμιά υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, διαβαθμίζουν ως απόρριτα έγγραφα για να μην τα δούμε εμείς. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Στη, στο Γερμανικό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί εκεί κάθε ε, βουλευτής ε, ε, ε διατηρεί απόρριτα έγγραφα και εκεί είναι πρόβλημα. Η συμφωνία πάντως δεν λειτουργεί έτσι όπως προβλέπεται από την ίδια τη συμφωνία. Η Κομισιόν αναφέρει ότι η συμφωνία έχει φτάσει σε επίπεδο ικανοποιητικό. Τι είναι αυτό το ικανοποιητικό. Χλιαρά πράγματα. Όχι καλά. Και αν οι συστάσεις που δόθηκαν στην πρώτη έκθεση, μετά την πρώτη έκθεση, γιατί υπήρχαν ακόμα ελλείψεις τώρα έχουν εφαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό, ε, αυτό σημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιε ελλείψει. Η συνεργασία της Europol με τη ΕΙΠΑ βελτιώθηκε μεν ω συνεργασία, αλλά αν βελτιώθηκε απλώ αυτό σημαίνει ότι εξακολουθούν και εκεί πάλι να υπάρχουν προβλήματα. Και για τους overseers, αυτούς επόπτες, την ευρωπαϊκή εποπτεία, αν πιστεύει η Κομισιόν ότι ο μηχανισμός αυτός ε, ε, λειτουργεί καλά. Αναρωτιέμαι τώρα, αυτό είναι θέμα πίστης ή υπάρχουν τεκμηρίωση, υπάρχει τεκμηρίωση ότι λειτουργεί η συνεργασία. Τώρα, η διαγραφή μετά από πέντε χρόνια τα είπαμε αυτά και εδώ υπάρχουν ακόμα προβλήματα από ό,τι φαίνεται. Τέλος, το θέμα της ε, συγκέντρωσης δεδομένων από ευρωπαϊκό έδαφος Μοιάζει όπως η συζήτηση στη Γερμανία για τα δημόσια κτίρια τα οποία κατασκευάζονται. Υπάρχει ένας προϋπολογισμός του κόστους και κατά τη διάρκεια γίνεται πιο ακριβό. Χτίζεται παρόλα αυτά, κατασκευάζεται το έργο, αλλά τρεπλασιάζεται το προπολογισμό του. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη εδώ συμφώνησαν σε ένα τέτοιο μοντέλο ε, συγκέντρωση δεδομένων από ευρωπαϊκό επίπεδο και είπαν ότι αν δεν γίνεται ε, άμα δεν λειτουργήσει δεν θα διαμαρτυρηθεί κανείς. Και άμα διαμαρτυρηθεί, παρόλα αυτά θα μείνουν τα πράγματα ως έχουν. Και θα σκεφτεί, και πρέπει να σκεφτεί το Κοινοβούλιο αν θα πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό να το δεχόμαστε, γιατί δεν είναι σωστό αυτό συμπεριφορά των κρατών μελών. Κυρία, η κυρία Ίνφελτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν μπορώ παρά να πηχήσω τα υποθέντα από τον κύριο Άλβαρο και την κυρία Σίπολ πάντα αστείο εγχείρημα η συζήτηση αυτή, διότι δεν γνωρίζουμε πράγματι τι συζητούμε. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες. Σημειώνω μόνο ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ αυτής της εκθέσεως και της ε, συνοπτικής εκθέσεως της τρισέλιδης που λάβαμε. Αν δεν έχουμε την πλήρη έκθεση δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Ίσως οι διαφορές μπορούν να εξηγηθούν από την επιτευχθήσα πρόοδο. Δεν το γνωρίζουμε όμως. Δεν ξέρουμε. Και είναι άκρος ανικανοποιητικό ότι δεν έχουμε το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 218 της συνθήκης να δώσουμε σύμφωνη γνώμη σε διεθνείς συμφωνίες. Σαν να υπογράφει κανείς ένα λευκό. Ε, συμφωνούμε και τίποτα άλλο. η προσεγγίση που ακολουθήσαμε για να καθησυχάσουμε τους εαυτούς μας όταν δεν μας άρεσε η συμφωνία, είπαμε θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγης τις εξέλιξεις. Αυτό εδώ δεν είναι ε, εκ του σύνεγγης παρακολούθηση. Ο Μιχλώδες το τοπίο. Ε, ο κ. Πρίμπελτ ίσως να έχει δίκιο, όλα να είναι υπέροχα και συμφωνία να είναι υπέροχη και φανταστική και ίσως όχι, δεν ξέρω. Δεν έχω τρόπο να το διαπιστώσω. όπως ανέφεραν και ο κύριος Αλβαρό και η κυρία Ζήπολ. Σίγουρα συμφώνησα με πάρα πολλούς μεγάλους δισταγμούς επ' αυτού, ε, θεωρώντας, δίνοντας, ε, θεωρώντας κατά τεκμήριον ε, αθώο τους την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόνο και μόνο γιατί μας υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εντός του έτους ένα σύστημα συλλογής στοιχείων θα είχε δημιουργηθεί δεν το καταλαβαίνω. Μιλάμε για λογισμικό, κάτι απλούστατο. Ε, γιατί γίνεται τόση φασάρια. Γιατί χρειάζεται τόσο χρόνο. Γιατί αντί απλού συστήματος συλλογής στοιχείων έχουμε επίσημη πρόταση για αυτό το ευρωπαϊκό TFTS που δεν το ζητήσαμε αυτό. Τώρα αποσύρθηκε η πρόταση από τη διάβαση στην εφημερίδα. Γιατί θέλαμε σύστημα για την ε, συλλογή στοιχείων εσείς επενείτε την χρήση των στοιχείων TFTP αν είναι τόσο υπέροχα γιατί δεν τα έχουμε τελικά. Ε. Τέλος. Υπάρχει και άλλη βάση δεδομένων τη είπα. Η TIDE. T-I-D-E. Που άλλαξαν οι οδηγίες που συλλέγει τα στοιχεία για περίπου 500.000 ανθρώπους που υπάρχουν λόγοι που ίσως τα αρχεία, τα στοιχεία θεωρείται ότι ίσως να περιέχουν ε, στοιχεία για τρομοκράτες. Δεν έχουν κατηγορηθεί επισήμως, δεν υπάρχουν επίσημες υπόνοιες. Αυτό αφορά Αμερικανούς πολίτες. Από τη δική μου εμπειρία η ΕΠΑ δεν αντιμετωπίζει καλύτερα τους μη Αμερικανούς πολίτες από τους Αμερικανούς. Θα με εξέπλητε λοιπόν αν αυτή η βάση δεδομένων έχει στοιχεία α, Αμερικανών πολιτών που δεν τους υποθέτονται για τίποτα. Και θα με εξέπλητε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για μη Αμερικανούς πολίτες, π.χ. Ευρωπαίους. Οι υποπτικές αρχές το έχουν επαληθεύσει, αν τα στοιχεία SWIFT, μήπως καταλήγουν τα στοιχεία SWIFT σε αυτή την βάση δεδομένων. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ακούσαμε ήδη. Κάποια συγκεκριμένα μόνο θέλω να αναφέρω από την έκθεση που λέει ότι η Europol από τον Ιούλιο του 2011 δεν έκανε άλλες, δεν διατύπωσε, δεν έστειλε άλλα αιτήματα, δεν ζήτησε άλλες πληροφορίες και είχε εγκρίνει όλες τις αιτήσει. Δηλαδή συνθηκολογεί. Συνθηκολογούμε μπροστά σε ένα σύστημα που δεν λειτουργεί και φαίνεται ότι η Europol δεν μπορεί καν να αποφασίζει και να ελέγχει αν ένα αίτημα πληρεί τις προϋποθέσεις της συμφωνίας και τις, ε, ε τους όρους της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή όχι και τα αιτήματα είναι έτσι διαμορφωμένα ώστε ουσιαστικά όλες οι πληροφορίες που έρεαν και πριν έτσι ρέουν και τώρα. Απλώς διατυπώνονται κάπως ιδιαίτερα τα αιτήματα για να υπάρχει έτσι, να μπορεί κανείς να τα ερμηνεύει όπως θέλει. Εγώ δεν καταλαβαίνω ποια δεδομένα διαβιβάζονται. Υποθέτω ότι διαβιβάζονται όλα τα δεδομένα. Εξακολουθούν να στέλνονται τα πάντα. Δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει αυτό, έτσι δεν είναι. Και θεωρώ ότι και το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, το Treasury Department λέει ότι τα περιτά δεδομένα ε, δεν... Ε, ε, ε, μπορούν να διαγραφούν μια φορά τον χρόνο. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται και δεν ξέρω, δηλαδή δεδομένα που δεν χρειάζονται πια, τι θα πει, άμεσα πρέπει να καταστρέφονται, όχι μετά από ένα χρόνο. Ε, επίσης, αυτή η συμφωνία, όπως την βιώνουμε και στην πραγματικότητα, δεν είναι τίποτα άλλο που επιβεβαίωση αυτού που βλέπαμε να είναι η πραγματικότητα και πριν. Και χειρότερα μάλιστα. Υπάρχει μια αλλαγή, ότι όλα αυτά γίνονται με, ε, ε, με το δικό μας πράσινο φως που το έχουμε δώσει. Αλλά δεν ε, συμφωνούν όλα αυτά με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εμείς ε, είχαμε ε, λάβει μια απόφαση από το Μάιο του 2010 και τώρα η συμφωνία παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό το είπε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, κατά του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την ε, διατήρηση δεδομένων με σκοπό τη διαβίβαση δεν είναι αυτή η χωρίς όρους διαβίβαση δεν συνάδει με την νομοθεσία, άρα η συμφωνία αντιβαίνει στην νοσιακή νομοθεσία. Ιδιαίτερα η πρακτική εφαρμογή της το αποδεικνύει αυτό. Και μάλιστα, και εγώ είχα συμφωνήσει, αλλά η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου τον Ιούνιο, όταν έγινε δεκτή η συμφωνία, είχε πει ότι αν ένα σύστημα συλλογής δεδομένων ε, ένα σύστημα, όχι σύστημα παρακολούθησης, σύστημα συλλογής αν δεν δημιουργηθεί, τότε μετά από πέντε χρόνια η συμφωνία αυτή θα πρέπει να τεθεί εκτός ισχύω. Και έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, θα παρακαλούσα να πάμε σιγά σιγά προς τα εκεί. Να αρχίσουμε δηλαδή την νομοθετική διαδικασία η οποία θα τερματίσει τη συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ. Η σειρά σας τώρα κύριε πρέπει να απαντήσετε. Ευχαριστώ πρόεδρε, δεν είμαι εδώ για να υπερασπίσω την DFTP. Απλώς μια έκθεση ήρθα να παρουσιάσω που προσπαθήσαμε να είναι αντικειμενική και νομίζω τα καταφέραμε. Και ευχαριστώ να δώσουμε λεπτομερείς πληροφορίες και φυσικά δεν θέλουμε να κρύψουμε τίποτα. Έτσι λοιπόν, ε, αυτό δεν είναι αστείο, είναι σκληρή δουλειά πολλών ανθρώπων για τρει μήνε. Αν το πετύχαμε αυτό, τότε κάναμε τη δουλειά μα. Ε, δηλαδή, ο στόχο του άρθρου 13 και τη σχετική αναθεώρηση δεν είναι να προετοιμάσει τι μελλοντικέ διαπραγματεύσει σε σχέση με, τη συμφων... την ε, συνέχιση ή με μη συνέχιση τη συμφωνία. Αλλά εγώ δεν έκρυψα τίποτα. πόσα λειτουργούν και πόσα δεν λειτουργούν τόσο καλά. Το συμπεράσμά μα είναι ότι η εφαρμογή είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, νομίζω, λέμε. Δηλαδή, ε, νομίζω ότι αν λέγαμε περισσότερα θα μας λέγατε ότι είμαστε προκατηλημένοι και περισπίζουμε ένα αμερικανικό μέσο. Λέμε λοιπόν πολύ ικανοποιητικοί. Και πολύ ικανοποιητικοί δεν είναι το ίδιο όπως ικανοποιητικοί. Υπάρχουν ε, κάποιες ελλείψεις, αλλά γενικά λειτουργεί αρκετά καλά. Τώρα, για το ένα θέμα, ε, το οποίο όντω εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια τη επανεξέταση, μία έλλειψη λοιπόν, είναι ο σημερινός ε, τρόπος ε, διαγραφής των δεδομένων ε, ουσιαστικά είναι προβληματικός γιατί δεν υπάρχει καθημερινή διαγραφή και λέει ότι το πολύ θα πρέπει να διατηρούνται πέντε έτη τα δεδομένα. Έτσι λοιπόν, αν δεν γίνεται η διαγραφή όπως πρέπει, αλλά σε κάποια στάδια, άπαξ το χρόνο ή δύο φορές το χρόνο, πρέπει να βρει κάποιο ένα σύστημα που να διασφαλίζει ότι δεν τηρούνται τα δεδομένα περισσότερο από πέντε έτη. Και εδώ το σημερινό σύστημα φαίνεται να λειτουργεί ως εξή ε, ότι θα πρέπει να διαγράφονται τα δεδομένα άνω των πέντε ετών παλαιότητας, αλλά αυτό δεν γίνεται έτσι λοιπόν, παραβιάζεται το σχετικό άρθρο της συμφωνίας. Και πάλι, είναι πολύ καλό που το εντοπίσαμε αυτό στην επανεξέταση και οι Αμερικανοί δύο εβδομάδες μόλις αργότερα επανήλθαν σε εμά και είπαν θα το αλλάξουμε αυτό. Και αυτό μας δείχνει ότι αυτές οι επαναθεωρήσεις έχουν κάποιο συγκεκριμένο αντίκτυπο και αυτό είναι καλό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μηχανισμό επαλήθευσης, άρθρο 4. Είναι λάθο, είναι απλά λάθος ε, και όλα τα μέλη της ομάδα ε, τη ε, αναθεώρηση το επιβεβαίωσαν. Η, το σχετικό άρθρο της GSP ήταν λάθος και αυτό το αναγνώρισαν όλα τα μέλη της ομάδας επαναξέτασης κατά τη διάρκεια της επαναξέτασης. Και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα δήλωση. Γι' αυτό εμείς στην ε, έκθεση συστήναμε να αποφευχθούν οποιασδήποτε παραπλανητικέ πληροφορίε στο κοινό όταν δεν είναι ορθές. Έτσι λοιπόν, ε, αυτό πρέπει να πούμε επί αυτού του θέματος, παραπληροφόρηση, που πιθανότατα μάλλον οφείλεται και σε έλλειψη συντονισμού από την πλευρά της GSP. Δηλαδή για το ποιος ε, εξετάζει τι και σε ποια χρονική στιγμή και μάλιστα αποφασίστηκε τον Οκτώβριο να γίνει μια τρίτη ε, επιθεώρηση από τις GSPR. Ε, η Κομισιόν βέβαια δεν είναι πολύ ικανοποιημένη με αυτό, αφού συζητήθηκε ε, για πολλές ώρες για το πώς λειτουργεί ο μηχανισμός της Europol και σε ποιο βαθμό θα πρέπει να εμπλακεί η GSP σε αυτό. Εγώ δεν θεώρησα ότι ήταν ε, πολύ ευτυχής η κατάσταση. Στη δική μου ομάδα επανεξέτασης να έχουμε δύο ανθρώπους που θα έπρεπε να επανεξετάσουν και τους αυτούς τους γιατί ήταν μέλη της GSP. Έτσι λοιπόν το πρόσημο ήταν ότι τα δύο μέλη της Επιτροπής Επανεξέτασης είχαν διοριστεί κατόπιν αιτήματος της Κομισιόν Δυνάμει τη ομάδα εργασία του άρθρου 29 και δεν θέλουμε να δώσουμε την εντύπωση ότι επιλέγουμε ε, κάποια μέλη τη ομάδα μας, αλλά αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα να το σκεφτούμε. Γιατί αν θέλετε αυτό μπορεί να, αποκαλυ... να αποκλειθεί, να... να αναφερθεί και ως σύγκρουση συμφερόντων. Τώρα για την πρόσβαση στα δεδομένα ε, συνεχίζονται οι συζητήσεις μεταξύ των αρχών προστασία δεδομένων της Επιτροπής ε, του άρθρου 29 και των Αμερικανικών αρχών για μια ομοιόμορφη διαδικασία για να αποφευθούν οποιασδήποτε παρεξηγήσεις. Αν θυμάμαι καλά, πριν δύο χρόνια ο μηχανισμός για να διαβαστούν αυτά τα αιτήματα μέσω των Εθνικών Αρχών Προστασίας των Δεδομένων είχε ζητηθεί ε, από αυτές τις αρχές προστασίας των δεδομένων στην Ευρώπη είχε ζητηθεί ένα πρόσθετο μηχανισμό. Χρειάζεται να καταρτιστούν οι άνθρωποι αυτοί για την DFTP. Αν χρειάζεται, ευχαρίστω να το κάνουμε. Μάλλον ε, δεν είναι συνήθι διαδικασία για αυτού. αλλά νομίζω ότι επιλύσαμε το πραγματικό πρόβλημα που είχαμε εκεί. Δηλαδή ότι μπορεί να ζητούσαν οι Αμερικανικέ Αρχέ πάρα πολλέ λεπτομέρειε ίσω για μια τέτοια πρόσβαση. Για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, σεβόμαστε τι δεσμεύσει μα. Δεν θέλω να επαναλάβω όσα είπε η στο Κοινοβούλιο και νομίζω όσα είπε και ο Γενικό Διευθυντή σε αυτήν την Επιτροπή πριν ε, λίγο καιρό. Κάναμε μια έκθεση που βάλαμε έκθεση, ένα έτος μετά τη θέση ισχύ και έχουμε μια ρήτρα στη συμφωνία και θα το πω στα γερμανικά γιατί το γερμανικό κείμενο λέει... Δυνατή εισαγωγή ενός ε, παρόμοιου συστήματος της Ένωσης. Είμαστε ανοιχτοί πάνω σε αυτό, είναι ανοιχτά τα αποτελέσματα. Κάνουμε μελέτη αντικτύπου που θα ολοκληρωθεί σε αρχές του επόμενου έτους και θα τηρήσουμε την προθεσμία των τριών ετών για να υποβάλουμε έκθεση. Αυτά κάνουμε λοιπόν εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα για το μηχανισμό υποπτίας. Εδώ έχουμε δύο δεδομένα. Όσα λέμε σε αυτή την έκθεση αναφέρονται σε δεδομένα, σε γεγονότα. Και πάλι πιστεύουμε ότι ο μηχανισμός αποπτίας λειτουργεί καλά σήμερα. Σελίδα είναι αυτό. Κατόπιν είχαμε κάποιε άλλε ερωτήσει. Νομίζω το άρθρο 4 το κάλυψα, Πρόεδρε. Χαίρομαι που μου στείλατε αυτό το άρθρο που εμφανίστηκε στις εφημερίδες και Αρχίζω να συνηθίζω πρόεδρε να έρχομαι εδώ για ένα θέμα και να με ρωτούν για άλλα θέματα, για την πρόσβαση σε έγγραφα, για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μία μέρα όταν ήρθα εδώ για τα PNR με ρώτησαν για το EPI. Τέλος πάντων, εμείς ε, ρωτήσαμε τις Αμερικανικές Αρχές και επειδή μιλάμε για την FTP, Θέσαμε την ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών και να σας πω τι λάβαμε ως απάντηση σήμερα ότι ε, το τμήμα της ε, καταπολέμησης χρηματοδότησης τρομοκρατίας ε, ε, παρουσιάζει κάποιες δικλίδες όπως κατέληξε, σύμφωνα με όσα κατέληξε, η έκθεση κομισιών, όλες τις δικλίδες παραμένουν σε ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα TFTP δεν ε, διασυνδέεται με άλλη βάση δεδομένων και δεν μπορούν να γίνουν αντίγραφα των δεδομένων και οι αναζητήσεις του TFTP μπορεί να γίνουν μόνο όταν υπάρχει αιτιολόγηση για τρομοκρατική πράξη. Και ε, οι επόπτες ε, ε, επιλέγονται από την Κομισιόν και από τις Αμερικανικές αρχές. Τώρα, το ουσιαστικό μήνυμα εδώ είναι ότι αυτό το σύστημα είναι stand-alone, λειτουργεί από μόνο του, δηλαδή δεν διασυνδέεται με άλλο σύστημα. Και από ό,τι καταλαβαίνω δεν συνδέεται όπως σας είπα με άλλο σύστημα και φυσικά Θα ρωτήσουμε τι Αμερικανικέ Αρχέ σε σχέση με τι πρόσφατε πληροφορίε που μα δώσατε και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρίμπε. Ξεπεράσαμε το χρόνο που είχαμε διαθέσει για αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη και είχαμε παρετηθεί από την ελπίδα να προλάβουμε και να συζητήσουμε τα σημεία του Συμβουλίου, αλλά βλέπω ότι υπάρχει προθυμία για συζήτηση. Αν μπορούμε να είστε σύντομοι θα βοηθήσει. Πολύ σύντομα λέει κύριε Εντφέλ, θέλω κάποιες διευκρινήσει. σω να παρεξήγησα και ελπίζω ότι παρεξήγησα. Ο κ. Πλήμπε νομίζω ότι είπε ότι ότι το συμπέρασμα ότι μεταφέρθηκαν στοιχεία από το JSP είναι ασφαλμένο το επιβεβαιώνεται. Ενδιαφέρον αυτό. Και μετά συνεχίζετε και είπατε ότι γι' αυτό επιλέξατε να μην αποκαλύψετε την έκθεση του JSP διότι δεν θέλετε να ενημερώσετε λανθασμένα με το κοινό. Η Ευρωπόλ μας είπε ότι ο λόγος για την μη αποκάλυψη έκθεση είναι διότι το ζήτησαν οι Αμερικανοί. Εξίσου κακός λόγος αυτός. Και φαίνεται υπάρχει διαφορά μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και JSP. Και λέτε ότι υπάρχουν άνθρωποι στην ομάδα που έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα. Αυτό είναι σοβαρότατες εικασίες. Θέλω να ακούσω περισσότερα γι' αυτό. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει τώρα, αλλά σίγουρα θα πρέπει γραπτώς να δοθούν διευκρινήσεις. Κύριε Πρίβε, μπορεί να μας βοηθήσετε να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Για να απαντή... Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι ναι κάποιες πληροφορίες στις στο ανακοινωθέντε τύπου για τη δεύτερη δική έκθεση ήταν εσφαλμένες πληροφορίες. Και το διευκρινίσαμε στην αναθεώρηση και όλοι συμφωνήσαν. Δεν θυμάμαι, αλλά ίσως γεράζω και ξεχνάω αυτά που είπα πριν από δύο λεπτά. Δεν θυμάμαι να σχολίασα το καθεστώς της εκθέσεως JSP και αν θα έπρεπε να εξεταστεί από μοτίμους ή όχι. Δεν είπα τίποτα πάνω σε αυτό. Βέβαια, Συμφωνώ με την άποψη της Ευρωπόλ μετά από τη δεύτερη έκθεση ε, των αρχών επιθεώρησης που γίνεται κάπως απειρχιωμένη, όπως έχουμε τη έκθεση, εμπεριέχει πράγματι συγκεκριμένα στοιχεία που έδωσαν οι Αμερικανικές αρχές υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πρέπει να αποκαλυφθούν άνευ συνένσεις των Αμερικανικών αρχών. Τι ήταν το άλλο, η άλλη ερώτηση. Α. Είναι απλά τα πράγματα. Επαναλαμβάνω. Όπως ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπόλ εκτέστα τα καθήκοντά της βάσει συμφωνίας, επαλήθευση του αιτήματο των Αμερικανικών αρχών και η εξέταση των ευρωπαϊκών αιτημάτων βάσει της ρήτρας αμοιβαιότητας και πώς οι πολιτικές αρχές ελέγχουν την Ευρωπόλ. Υπήρχαν αμφισβητήσεις από πλευράς Αμερικανών όσο φορά αυτό. Διότι το Δικαιωτικό Συμβούλιο και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων ελέγχει την Ευρωπόλ. Ο τρόπος αντιμετώπισης διενέργειας των ελέγχων επίσης ήταν θέμα βασικό των συζητήσεων για την φετινή αναθεώρηση και θεωρώ κάπως ατυχές ότι στην ομάδα αναθεώρησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως υπάρχουν δύο άτομα που είναι επίσης μέλη αυτού του οργανισμού που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα στην αναθεώρηση. Πώς αυτοί μπορούν λοιπόν να κινηθούν χωρίς να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων, ε, τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν παρά να αυτά που έκαναν σε άλλο φορέα. Αφελώς σκέπτομαι, δεν είμαι εμπειρογνώμων, δεν ανήκω στην Όλαφ, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι που ίσως να οδηγεί ε, ενδεχομένω σύγκρουση συμφερόντων. Ευχαριστώ. Αυτά για την ώρα. Σα ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και μοιραστήκατε μαζί μας την όλη κατάσταση όσον αφορά το ευαίσθητο αυτό θέμα. Όπως και πριν με την Επίτροπο Ρέντινγκ, δρατώμεθα της ευκαιρίας και με εσάς να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τις χριστουγεννιάτικες διακόπες, για τις γιορτές. Ευχαριστώ. Now, move on. As... Προχωρούμε. Πάμε στο σημείο που αφορά το ζήτημα που επεξεργάζεται το, ο κύριος Ντεμέρα είπαμε ότι αναβάλλεται και πάμε στο σημείο 18, έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Δεύτερη έκθεση όσον αφορά τη λειτουργία της, του, χώρου Σέγγεν, Μάιος 2012 με Οκτώβριο 2012. Δύο φορές το χρόνο δημοσιεύει αυτή την έκθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν και μπορούμε να ανταλλάξουμε επί τη ευκαιρία απόψεις. Θα δώσω το λόγο στην ε, κυρία Μπελίντα Πάικ που είναι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά θα ξεκινήσει τη συζήτηση. Κυρία Πάικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ να παρουσιάσω τη δεύτερη έκθεση. Ήρθα εδώ και πριν τις καλοκαιρινές διακοπές να παρουσιάσω την πρώτη έκθεση. Όπως ξέρετε, η Κομισιόν θεωρεί σημαντικό το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να έχουν την ευκαιρία σε τακτική βάση να εξετάζουν τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν και να αποτιμούν τις εξελίξεις ε, μέσα σε 6 μήνες και επίσης να δίνουν πολιτική καθοδήγηση για τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν. Η έκθεση αυτή συζητήθηκε στο Συμβούλιο ΔΕΗ στις 6 Δεκεμβρίου και θα ήθελα πολύ γρήγορα να συνοψίσω κάποια τα κύρια σημεία, καταρχήν για τα εξωτερικά σύνορα, κατόπιν για τα εσωτερικά, για τη διεύρυνση και τις θεωρήσεις. Καταρχήν για τα εξωτερικά σύνορα παραμένουν υψηλέ οι πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, κυρίως σε, ε, ε, σε κάποια hot spot, κυρίως στα χρυσά σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, ε, αλλά νομίζω ότι μπορούμε με χαρά να σημειώσουμε ότι οι αυξημένε προσπάθειε των ελληνικών αρχών στο να ελέγξουν αυτό το σύνορο οδήγησαν σε σημαντική μείωση στον αριθμό των παράτυπων διελεύσεων σε αυτόν τον τομέα. Βέβαια η κατάσταση στη Συρία μα ανησυχεί ιδιαίτερα, υπάρχει και το θέμα τη ανθρωπιστική βοήθεια, Πέραν αυτού η Κομισιόν αναπτύσσει ένα πρόγραμμα προστασία στι γειτονικέ χώρε. Ο στόχο είναι να διασφαλίσουμε ότι νομιμοποιείται η παρουσία τη και το καθεστώτο δεν μπερδεύεται όπω αυτό το παράτυπο μεταναστών. Ταυτόχρονα λαμβάνουμε κάποιε εκθέσει για κάποιου κάποιου μετανάστε που πνίγονται ε, στη Μεσόγειο και ιδίω ε, στο Αιγαίο, όπως ακούσαμε πρόσφατα. Επομένω, ε, καλωσορίζουμε τι διαπραγματεύσει για να δημιουργηθεί η Eurosur, καθώ αυτό το σύστημα θα περιορίσει την απολύτω ζωή στη θάλασσα. Και επιπλέον, όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση του Συμβουλίου που κανόνε κανόνες και κατευθύριες γραμμές ε, για ε, τις επιχειρήσεις της Frontex ε, στα θαλάσσια σύνορα. Πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των επιχειρησιών μας. Το Δικαστήριο δέχτηκε ότι η απόφαση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να υιοθετηθεί μια νέα απόφαση και η Κομισιόν σχεδιάζει να παρουσιάσει νομοθετική πρόταση στις αρχές του 2013 για να αντικαταστήσει την απόφαση του Συμβουλίου. Για τα εσωτερικά σύνορα τώρα συνεχίζουμε να λαμβάνουμε καταγγελίες από τους πολίτες ε, σε ό,τι αφορά ε, τους, ότι υπάρχουν έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα και τερευνούμε αυτά σοβαρά. Κάποιες καταγγελίες φαίνεται να είναι σταθερές, αλλά νομίζω ότι όλοι πρέπει να επαγρυπνούμε για οτιδήποτε μοιάζει με ελέγχους στα σύνορα, σε εσωτερικά σύνορα ή σε εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία στα εσωτερικά σύνορα. Και όπως ξέρετε, τα κράτη-μέλη υπό κάποιε προποθέσει σε προσωρινή βάση έχουν τη δυνατότητα να επανεισάγουν ελέγχου στα ιστορικά του σύνορα και όπω ε, αναφέρεται στην έκθεση, δύο κράτη-μέλη το έπραξαν αυτό στο εξάμεινο που καλύπτεται την έκθεση Ισπανία και Πολωνία και καθώς η περίοδος, από μάλλον από την περίοδο αυτή είχαμε μία νέα κοινοποίηση από την Ορβηγία ότι υπήρξε ε, του μέτρου όταν απονομήθηκαν τα βραβεία Νόμπελ. Τώρα εξηγούμε στην έκθεση τα σημαντικά μέτρα που έχουν ελευθεί για ε, να επιτευχθεί ένα σημαντικό στόχο και η Κομισιόν θεωρεί ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία ε, πληρούν όλου τους στόχους, ε, σέβονται το κεκτημένο Σέγγεν και καλωσορίζουμε το να λάβει το Συμβούλιο θετική απόφαση για την προσχώρηση Ρουμανίας και Βουλγαρίας στη Σέγγεν. Και τέλος ε, η έκθεση καλύπτει ορισμένα θέματα για την πολιτική θεωρήσεων και ιδίω να τονίσω ότι το VIS ε, έχει τώρα καλύψει δύο νέες περιοχές ανατολικά και συνεχίζει να λειτουργεί καλά. Πιστεύω να βρείτε την έκθεση αυτή χρήσιμη. Περιμένουμε τα σχόλιά σα ε, για την έκθεση αυτή και για θέματα που θα θέλετε ίσω να εμβαθύνουμε σε μελλοντικέ εκθέσει. Θα συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε τι εκθέσει αυτέ κατά εξάμεινο και ελπίζουμε να σα βοηθούν στον προβληματισμό σα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πάη εκ μέρου τη Κομισιόν. Σα ευχαριστούμε για την αφοσίωσή σα και για τη δέσμευσή σα ε, για το φάκελο αυτό. Αν ε, και όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι η καλύτερη χρονική στιγμή να συζητηθεί τώρα, καθώς έχει περάσει και η ώρα. Αλλά να δώσουμε το λόγο σε όσους παραμένουν στην αίθουσα. Κύριε Παπα-Νικολάου, το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δεύτερη έκθεση που αφορά το χώρο Σέγγεν. Άκου, ε, διάβασα την έκθεση και παρατήρησα ότι η έκθεση αυτή ξεκινά με περιγραφή όσων συμβαίνουν στα εξωτερικά σύνορα και κυρίως στα ελληνοτουρκικά σύνορα και πώς γίνονται βελτιώσεις και ποιες είναι οι θετικές εξελίξεις. Στην πρώτη έκθεση υπήρχαν πολλές επικρίσεις στα σχόλια που αφορούσαν την κατάσταση σε αυτή την περιοχή και τις προσπάθειες της Ελλάδας που χρειαζόταν. Τώρα είναι το αντίθετο που αναφέρεται, θετικές εκδηλώσεις και 1.800 αστυνομικοί πήγαν στα σύνορα και πετύχαμε έτσι μεγάλες βελτιώσεις όσον αφορά τα αποτελέσματα και την μείωση των μεταναστευτικών ροών, όσον αφορά τους παράνομους μετανάστες. Ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φρονεί ότι αυτή η κατάσταση θα γίνει μόνιμη για το εγγύς μέλλον, διότι ξέρω ότι αυτές οι προσπάθειες απέτησαν σημαντικές ε, χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νέα υποδομή, τεχνική υποστήριξη από τη Frontex, και ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλα Μέχρι τώρα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω δράση στο εγγύς μέλλον. Πιστεύετε ότι αυτή η εξέλιξη θα είναι σταθερή και δεν θα αλλάξει μέχρι την επόμενη έκθεση. Σας ευχαριστώ. Η ε, κυρία Τσίπελ. Και εσείς μια ερώτηση γρήγορη. Πολύ σύντομα μια παρατήρηση σε ένα άλλο σημείο της ημερήσιας διάταξης σήμερα είπαμε ότι υπάρχει ένας μηχανισμός στις υποψήφιες χώρες εις ό,τι αφορά τα κριτήρια της Κοπενχάγης αλλά αυτά δεν τα εξετάζουμε αν ισχύουν και εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Και στο θέμα του χώρου του Σέγγεν, καλό είναι να στρέψουμε την προσοχή μας όχι μόνο στα εξωτερικά σύνορα, αλλά να δούμε πολύ συγκεκριμένα τι γίνεται και στα εσωτερικά σύνορα. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια Είχαμε κάποιες αναφορές και τόπικοι κομισιόν που έδειχναν προβλήματα στα εσωτερικά μας σύνορα. Και νομίζω ότι και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί στη συζήτηση έτσι όπως ε, προβάλλεται γίνονται συζητήσεις για τα εξωτερικά, όχι όμως και για τα εσωτερικά σύνορα. Μην τα ξεχνάμε. Ευχαριστούμε. Κυρία Πάεκ, θέλετε να δευτερολογήσετε μετά από αυτά που ακούσατε από τα μέλη. Ευχαριστώ λέει κυρία Πάικ. Ναι, πράγματι με τα χαράς ε, σημειώνουμε τις βελτιώσεις τους τελευταίους μήνες όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά χεσαία σύνορα και πρέπει να ξέρουμε ότι βέβαια, όχι βέβαια, δεν είναι έκπληξη ότι υπήρξε αλλαγή των μεταστατικών ροών και μάλιστα λόγω της αστεριότητας εκείνων που διακινούν τους μετανάστες και αυτού που παρέχουν διευκολύνσεις. Υπήρχε μετακίνηση προς τα θαλάσσια σύνορα με τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Είδαμε την τραγωδία που συνέβη προσφάτα στη Λέσβο. Και γι' αυτό ε, απευθύνεται το Κοινοβούλιο γρήγορα κονδύλια και τελικά ασκείται επιχείρηση Ποσειδών στην περιοχή Ελπίζουμε ότι θα διατηρηθούν οι επιτευχθείς πρόοδοι, αλλά η προσωρινή μετάθεση ε, συνοριοφυλάκων στα σύνορα πρέπει να ενισχυθεί και να γίνει πιο βιώσιμη, πιο διαρκής και συνεχίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές όσον αφορά ολοκληρωμένη πολιτική διαχείριση των σύνορων χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες διαθέσιμες τεχνικές. Εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι μπορούν να απορροφήσουν τη διαθέσιμη χρηματοδότηση από το Ταμείο για τα Εξωτερικά Σύνορα. Υπάρχει πρόβλημα στον αφορά τη χρηματοδότηση, το αναγνωρίζουμε και ήταν ένα θέμα το οποίο ε, το συζητεί το Κοινοβούλιο και ελπίζουμε τώρα και το Συμβούλιο θα συζητήσει, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό τη χρηματοδοτήσεω. Ελπίζω, αλλά δεν μπορώ να υποσχεθώ, ελπίζω ότι στην επόμενη έκθεση θα μπορούμε να δείξουμε ότι η βελτίωση αυτή διατηρήθηκε όπως ε, υπενόησε το αξιότιμο μέλος. Είναι σημαντική πρόοδος, δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη όμως ότι ίσως μπορεί να υπάρχει επαναχώρηση, αλλά χρειάζεται στενή συνεργασία από αυτού και βέβαια να δούμε ποιος είναι και ο ρόλος της Frontex και πολύ σημαντική συνεισφορά από τα κράτη-μέλη προς τις κοινέ επιχειρήσεις Frontex, Αταλάντα και ε, στη, συγγνώμη, στα χερσαία σύνορα και στα θαλάσσια να η, η έλλειψη εσωτερικών συνόρων σημαντικότατο θέμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και θα είναι σημαντικό στοιχείο όσον αφορά την αξιολόγηση του μηχανισμού Σέγγεν. Ξέρω ότι η τριμερής διάλογος συνεχίζεται μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι επίσης εξασφαλίζουμε απουσία ελέγχων στα εσωτερικά ε, σύνορα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πάικ. Άλλη ερώτηση, άλλο σχόλιο υπάρχει από τα μέλη μας. Εάν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, σας ευχαριστούμε κυρία Πάικ για την παρουσίαση και ο Πρόεδρος δράτε της ευκαιρίας να διαβιβάσει ένα μήνυμα καλής βούλησης, καλής θέλησης προς τα μέλη, τα μέλη της γραμματείας, μάλλον ευχές. Γραμματεία προσπαϊσταμένος και στους διερμηνείς και τον ευχαριστούμε γι' αυτό που ε, δούλεψαν και εξυπηρετούν τόσο καλά αυτό το νίκο της πολυγλωσσίας του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές ευχές όχι μόνο για τις χριστιανιάτικες διακοπές, για τις γιορτές, αλλά και για τον καινούριο χρόνο, το 2013, ευχόμαστε όλοι το νέο έτος να ρίξει φως, να δείξει ότι υπάρχει φως στο τέλος της σύραγγας αυτής της ατέρμονος ε, ε, που μας έκανε υποφέρουμε τόσο πολύ και έθεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δεινή ε, κατάσταση, σε μεγάλη πίεση επί μακρόν. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους και θα συνεχίσουμε τις εργασίες Επιτροπής Ελευθεριών στις 10 Ιανουαρίου στις 9 το πρωί. Μέχρι τότε περάστε ε, καλά, καλά Χριστούγεννα και ένα πολύ ευτυχισμένο καινούριο χρόνο σας εύχομαι.